Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ πολύ. Η κυρία Γεωργίεβα θα φτάσει σε τρία περίπου λεπτά. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίρρηση για τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Τα επόμενα λοιπόν λεπτά θα φτάσει εδώ η κυρία Γεωργίευα, η Επίτροπος, η οποία θα μας παρουσιάσει το σχέδιο αναθεώρησης και ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές, του δύο συνεισηγητές όσον αφορά το σχέδιο ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου στον μόνιμο εισηγητή μας έπειτα για τον δημοσιονομικό κανονισμό, στον μόνιμο εισηγητή για τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Στη συνέχεια, στον σκιώδη εισηγητή όσον αφορά το σχέδιο αναθεώρησης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και στη συνέχεια στους συντονιστές. Έχουμε όμω ήδη καθυστερήσει και ξέρετε ότι έχει πάρα πολλές συνειδημένες υποχρεώσεις η κυρία Γεωργίευα. Προκειμένου λοιπόν είναι σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας, θα σας πρότεινα τα τρία λεπτά τα οποία προβλέπονται για τις δικές σας τις αγορεύσεις να μειωθούν σε δύο λεπτά. Διότι διαφορετικά η κυρία Γεωργίευα θα χρειαστεί να αποχωρήσει χωρίς να καταφέρει να απαντήσει στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Συνεπώς, αν συμφωνείτε, θα μιλήσει ο καθένας δύο λεπτά και εκ των προτέρων σα ζητώ κατανόηση για τον περιορισμό που επιβάλλω στον χρόνο αγόρευσης. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα τελειώσει και το suspense, περιμένουμε αλλά δεν θα ολοκληρωθεί το όνειρό μας. Χθε, στη συζήτηση που έγινε για το σχέδιο προπολογισμού για το έτος 2017, είπα ότι ακόμα ονειρευόμαστε. Ότι α, σήμερα το πρωί θα ακούγαμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι οι προτάσεις που θα μας έκανε ουσιαστικά θα ενίσχυαν, θα εμπλούτιζαν το όνειρο αυτό και ότι στη συνέχεια θα ερχόταν και η κυρία Γεωργίευα με το σχέδιο αυτό ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να τροφοδοτήσει και αυτή περισσότερο και να εμπλουτίσει αυτό το όνειρο, αυτό το ιδεώδε. Α περιμένουμε λοιπόν λίγο ακόμα. Νομίζω ότι οι συνεργάτε τη Επιτρόπου φτάνουν και ναι, ναι, βλέπω την κυρία Γεωργίευα. Α τη χειροκροτήσουμε. Κυρία Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Με ιδιαίτερη ανυπομονησία καταλαβαίνετε ότι ε, περιμένουμε να σας ακούσουμε και όσοι ήμασταν παρόντες ε, στα τέλη του 2013 όταν πρωτοεγκρίθηκε το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 τότε Πολλοί από εμά χρεσήκαμε να κάνουμε κάποιες θυσίε και θέσαμε δύο προποθέσει. Πρώτον, να δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλού επίπεδου που θα επεξεργαζόταν ε, τις, ε, πιθανού ε, πιθανούς δυνατούς ιδίους πόρους στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακούσαμε και μια παρουσίαση από τον Μάριο Μόντι την προηγούμενη εβδομάδα και πρέπει να περιμένουμε όμως ακόμα και να ακούσουμε και νέες προτάσεις προκειμένου να έχει νέους ίδιους πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε πει επίσης τότε, είχαμε θέσει ως δεύτερη προϋπόθεση την ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ελπίζαμε λοιπόν τότε και ελπίζουμε ακόμα ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και σας δίνω ευθύ αμέσως το λόγο κυρία Γεωργίευα και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε για αυτή την καθυστέρηση. Έπρεπε να γίνει μια συνέντευξη τύπου με τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν και την είπατε εκπρόσωπο Μογκερίνη και έπρεπε να απαντήσω μια ερώτηση πρωτού έρθω εδώ. Ε, συγγνώμη λοιπόν, βαθιά συγγνώμη. Είπατε ότι θέλετε να κρατήσει το όνειρό σας. Και χαίρομαι που είπατε τα πράγματα λίγο λιγότερο αισιόδοξο από ό,τι θα μπορούσατε. Το όνειρό μας να γίνει πραγματικότητα. Το όνειρο λοιπόν πιστεύω ότι θα κρατήσει και μπορούμε να δουλέψουμε μαζί για να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε εργαστεί τους τελευταίους μήνες πολύ εντατικά για την ενδιάμεση αναθεώρηση και την πρόταση αυτή για αναθεώρηση που θα σας υποβάλω και αναγνωρίζω πραγματικά το έργο αυτής της Επιτροπής και πολλών άλλων στο Ευρωκοινοβούλιο φρόντισαν να υποβάλουν ιδέες, συστάσεις, ενδείξεις. Το ίδιο και οι Υπουργοί του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ, που δύο φορές μου έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε. Και το ίδιο και για τους συνεργάτες μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκαν σκληρά για να έχουμε μια πρόταση που να είναι ουσιαστική, διεξοδική και δίκαιη. Να ξεκινήσω από το πακέτο, τη δέσμη μέτρων τρεις συνιστώσεις ε, ε, περιλαμβάνει το έγγραφο εργασίας και ε, την, ανακεφαλαίωση της προτινόμενης μεταρρύθμισης, την ευελιξία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την προτάση απλούστευσης των κανόνων εφαρμογής των δημοσιονομικών κανονισμών και των λεγόμενων εφαρμοστικών πράξεων Omnibus. Έχουμε και κάποιες συνδεόμενες πράξεις, τρεις θέλω να τονίσω, οι οποίες είναι εμβληματικές για μας. Τη μία για το επενδυτικό πρόγραμμα μέχρι το 2020, το ΕΦΣΥ, για να έχουμε διπλάσιο μέγεθος από ό,τι τώρα, δηλαδή να φτάσουμε τα 500 εκατομμύρια, μια πρόταση για ένα νέο ταμείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις εξωτερικές επενδύσεις μας δηλαδή, και μικρότερες σε μέγεθος προτάσεις αλλά νομίζω ότι θα σας αρέσουν εσάς ιδιαιτέρως, δηλαδή στο δημόσιο πεδίο, οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ελεύθερο δωρεάν Wi-Fi διαδίκτυο. Εδώ λοιπόν να δούμε το πλαίσιο εντός του οποίου θα ε, προχωρήσει αυτή η πρόταση. Τα γνωρίζετε πολύ καλά διότι μου έχετε ήδη δώσει κάποιες από τις ε, αντιδράσεις σας ένας νέος προπολογισμό, ο οποίος να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα. Η δυνατότητά μα να καθορίσουμε σαφώς πού δαπανούμε, πού δαπανούμε πώς, δα, πώς δαπανούμε και πώς αποτιμούμε τις δαπάνες Δηλαδή, να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Επίση, το πώς προβάλλουμε τις ενεργές μας στους πολίτες Αυτό είναι προφανώς ένα θέμα άκρος σημαντικό για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα επικριτικά σχόλια. Λαμβάνουμε βήματα και υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Να σας θυμίσω ότι τις 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη δεύτερη συνομιλία, διάσκεψη για να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα του προπολογισμού και υπολογίζω στην εργή σας συμμετοχή σε αυτή. Εάν δείτε τη δέσμη μέτρων που προτείνουμε, υπάρχουν τρεις σαφείς στόχοι. Να προβλέψουμε τους πόρους και τα κονδύλια στους τομείς προτεραιότητας, που είναι σαφείς, εργασία, ανάπτυξη από τη μία, ασφάλεια, μετανάστευση, πρόσφυγες, εξωτερικά σύνορα από την άλλη. Δεύτερον, να κάνουμε και να δώσουμε συνέχεια σε όσα ξεκινήσατε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη κινητικότητα στον προπολογισμό και τρίτον μείωση του γραφειοκρατικού άρθρου Λιγότεροι κανόνες που, ε, με ε, εξάλληψη των περιτών που δεν έχουν καμιά προστιθέμενη αξία. Εάν δούμε από δημοσιονομική σκοπιά το πακέτο, έχουμε 12,8 δις, εκ των οποίων η ενδιάμεση αναθεώρηση προβλέπει 6,3 δις κονδύλια από αυτή τη στιγμή δεν έχουν δεσμευτεί και θα στοχευθούν, θα κατευθυνθούν προς τις ε, κορυφές μας προτεραιότητες. Τεχνική προσαρμογή της συνοχής, κάτι που ήδη γίνεται, 5,6 δις και επιπλέον δαπάνες για τη μετανάστευση. Κάτι που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς το σχέδιο του προπολογισμού το 2017 1,8 δις. Εάν δείτε τα 6,3 δις, νέο στοιχείο για σας αυτό, κατανέμονται 2,4 για τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, 3,9 δις για τη μετανάστευση και έχουμε εφαρμόσει αυστηρότατους κανόνες για τους επιμέρους στόχους. Ενίσχυση των προγραμμάτων που δίνουν αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Στο Κοινοβούλιο γνωρίζω ότι τα στηρίζονται τα προγράμματα αυτά. Το COSME 200 εκατομμύρια, το Horizon 2020 400 εκατομμύρια, η διασύνδεση της Ευρώπης στις μεταφορές 400 εκατομμύρια και το Erasmus Sin 200 εκατομμύρια. Αυτά είναι προγράμματα με τεράστια ζήτηση και υπάρχουν ενδείξεις και βεβαιότητα ότι θα δώσουν αποτελέσματα. Προσθέτουμε ένα δις για την πρωτοβουλία προσχόλησης των νέων και ένα δις από το κοινωνικό ταμείο θα προσθεθεί σε αυτό. Να υπογραμμίσω ότι ενθαρρύνουμε τις τρεις χώρες που είναι μεγαλύτεροι δικαιούχοι της τεχνικής προσαρμογής στη συνοχή, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, και που τυχαίνει να είναι χώρες με σοβαρότατα προβλήματα στην ανεργία των νέων να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο που ενισχύει για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Μπορεί να θελήσουν να το χρησιμοποιήσουν για τη μετανάστευση. Μπορεί, υπάρχουν χώρες, εάν σκεφτώ την Ιταλία και την Ελλάδα δηλαδή, ε, έχουν σοβαρότατα προβλήματα και σε αυτό το τομέα. και κάναμε, για πέρσι, και κάναμε κάποια πράγματα που μα τα έχει ζητήσει έτσι και στο Κοινοβούλιο. Να μειώσουμε την εγγύηση από 50% σε 35%. Οι βουλευτέ όταν το άκουσαν μα είπαν σα το είχαμε πει. Εγώ εδώ πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζαμε. Δεν γνωρίζαμε πώ θα λειτουργήσει η εγγύηση. Τώρα γνωρίζουμε και μπορούμε να έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση και να είμαστε κάπω λιγότερο επιφυλακτικοί. Και μετά 50 εκατομμύρια με το WiFi για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σκέλος της μετανάστευσης, δύο, μεγάλες, ε, δύο μεγάλα σύνολα, εξωτερική δράση, Frontex ε, και ο νέος οργανισμός και άλλες δράσεις για να απορροφηθεί, να αντιμετωπιστεί η πίεση από την κρίση και έπειτα εξωτερική δράση για να δούμε τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης 1,4 δις. Βλέπετε ότι αυτό κατανέμεται σε 250 ε, εξωτερικό ταμείο επενδύσεων, έπειτα τα σύμφωνα μετανάστευση 750 εκατομμύρια και 385 για την δυνατότητά μας να περάσουμε σε εξωτερική δράση από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με την μακροοικονομική δημοσιονομική στήριξη. Αυτό είναι ένα χαρτοφυλάκιο κονδυλίων. Αυτή είναι η συλλογιστική. Ποια προγράμματα δίνουν αποτελέσματα. Ένα. Δύο. Νέο χρήμα για δράσει που πιστεύουμε ότι θα έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία. Κατά δεύτερον, αυξάνουμε την ευελιξία και κινητικότητα. Την ευκαμψία να τονίσω ότι εδώ χρειαζόμαστε ομοφωνία στο Συμβούλιο για να συμφωνήσουμε. Για το διπλασιασμό του μεγέθους, του υπάρχοντος εργαλείου ευελεξίας και του Ταμείου για την εμετώπιση Κατεπηγόντων από τα 500 εκατομμύρια στο 1 δις, από 250 δηλαδή σε 500 εκατομμύρια. Για να δημιουργήσουμε και εδώ αυτό είναι η ιδέα του Κοινοβουλίου και την έχουμε ακολουθήσει και την έχουμε υιοθετήσει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, δεσμεύσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουμε ένα ταμείο ε, έκτακτης ανάγκης για τις κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι όταν ξεσπάει μια κρίση πρέπει να ε, ενεργοποιηθούμε αμέσως. Είναι λοιπόν καλή ιδέα να πάρουμε ποσά που δεν έχουν ταπανηθεί για να δημιουργήσουμε αυτό το ταμείο. Θέλουμε στην εξωτερική δράση μας να είμαστε πιο επιφυλακτικοί στις ε, πρώτερες δεσμεύσεις μας, με το 10% ως ένα μαξιλαράκι ευελιξίας εκεί, αλλά ταυτόχρονα στο συνολικό περιθώριο για τις, δεσμεύσεις, για τις δεσμεύσεις δεν θέλουμε να υπάρχει ε, τόσο μεγάλος περιορισμός. Θέλουμε να άρουμε το, το εμπόδιο εκεί. Έπειτα, οι προβλέψεις για τις τρέχουσες πληρωμές. Εδώ αυτό που βλέπετε όλοι το 2016 και το 2017 δυστυχώς είμαστε πολύ ε, κάτω από το προβλεπόμενο επίπεδο. Δηλαδή οι λογαριασμοί θα φτάνουν στη, στην πόρτα μας ε, πολύ καθυστερημένα. Στη Βουλγαρία ήδη μου τηλεφωνούν και μου λένε ότι ανησυχούν πολύ με τον προπολογισμό το 2017. Τι σημαίνει μου λένε, θα έχουμε λιγότερα χρήματα. Η απάντηση είναι όχι. Απλώς σημαίνει ότι θα έχετε λιγότερους λογαριασμούς να, να πληρωθούν ε, που θα φτάνουν στο γραφείο μας όμως. Ε, δεν θα έχετε λιγότερα χρήματα, αλλά φέτος δεν πληρώνουμε τόσους λογαριασμούς όσο θα θέλαμε και αυτό δυστυχώς δεν θα λυθεί πολύ γρήγορα. Και εκτός και αν κινητοποιηθούν όλοι εντατικά γι' αυτό, θα παραμείνουμε ε, στο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει και ο κύριος Ντεπρέ. Τώρα, ε, τα ανώτερα όρια των πληρωμών, οροφές, θα είναι βιώσιμα οι στόχοι μας εάν οι πληρωμές για τα ειδικά εργαλεία υπολογιστούν πάνω από τα ανώτατα όρια. Ξέρετε ότι αυτό το ζήτημα ακόμα απομένει να επιληθεί μεταξύ ε, ημών και του Συμβουλίου. Το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές αξιοποιείται πλήρω για να προβλέψουμε τη μέγιστη απαιτούμενη ευελιξία. Και αυτό πάλι είναι κάτι που πρέπει να το επεξεργαστούμε. Μιλάμε εδώ για σημαντικά ποσά με ε, τα ειδικά εργαλεία που μπορεί να βρεθούν σε μια κλίμακα από 10 δις, ήδη έχουμε 3,4 δις που έχουν ε, προβλεφθεί, έχουν εκταμιευθεί κάποια είδη εκ των προτέρων. Δεν είναι απλό το ζήτημα και δεν θα είναι και εύκολο να επιληθεί. Οι συνολικές μας προβλέψεις, αν δείτε τώρα τις προβλέψεις τα και πριν, πρέπει να είναι πάνω από τις οροφές. Ιδάλλως, θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Ήδη έχουμε εναντικοποιήσει πληρωμές για το 2017 στην πρόταση για το 2017 δεν ε, έχουμε όμω καλύψει όλα αυτά που έπρεπε να έχουν ε, εκταμιευθεί για το 2017. 350 εκατομμύρια από την απόφαση του 2014 δεν έχουν ε, ενεργοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στην περίοδο όπου θα έχουμε βάλει τα ποσά πάνω από τα ανώτατα όρια εγκαίρως, διότι αλλιώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα προηγούμενα προβλήματα. Τώρα, για τους κανόνες δαπάνης και την απλούστευσή τους. Δύο πράγματα. Ένα ενιαίο ε, σύνολο κανόνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούν να ε, κάνουν ε, οι αρμόδιοι φορείς την, τον έλεγχο με τις δικέ του δυνατότητε, Δηλαδή να δείξουμε εμπιστοσύνη στις υπάρχοντες ανθρώπινους πόρου παρά να κάνουμε επικάλυψη των ίδιων ε, δραστηριοτήτων. Και έπειτα και απλούστευση των 25 νομοθετικών πράξεων οι συνάδελφοί μα στοχεύουν σε ένα ε, εγχειρίδιο που να είναι το 1 τέταρτο του σημερινού στο, στην εκτασή του. Ο, το σύνολο των δημοσιονομικών κανόνων, το θέμα αυτό σχετίζεται άμεσα με την ενδιάμεση αναθεώρηση, όμως υπάρχουν κάποια σκέλη που θα τα δούμε εκ των υστέρων. Θα είναι σημαντική νομοθετική δουλειά που θα έχουμε να κάνουμε, αλλά αυτό που θέλουμε να δούμε δεν είναι απλώς απλουστευμένοι κανόνες. Θέλουμε αποτελεσματικότερο συνδυασμό των εργαλείων. Θέλουμε να δούμε υποβολή εκθέσεων που να βασίζεται και να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και πολύ σημαντικό για μας, θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Θέλουμε οι άνθρωποι μας να έχουν λέγειν στο τι θέλουν ο ευρωπαϊκός προπολογισμός να τους προσφέρει. Ένα παράδειγμα του Wi-Fi for EU. Wi-Fi για όλους. Γιατί να μην μπορούν οι πολίτε να υποφελούνται από το δωρεάν WiFi ασχέτω που θα βρίσκονται τα hot spots, του τριοδρομικού σταθμού, σε βιβλιοθήκε ή στην κεντρική πλατεία. Αλλά το να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν συμμετοχή ώστε να αισθάνονται ότι του αφορά, του ανήκει ο προπολογισμό περισσότερο από ό,τι σήμερα είναι σημαντικό. Το ίδιο με τον πολύ απλό κανόνα. Περισσότερο, περισσότερη διαφάνεια στον προπολογισμό σημαίνει και περισσότερη λογοδοσία. Δηλαδή η λογοδοσία δεν βαρύνει πλέον ως ευθύνη τόσο πολύ τους ε, ελεγκτές μόνον, αλλά και τους πολίτες μας. Και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ σε αυτή τη διαφάνεια, διότι ήδη μίλησα πολύ ώρα. Το μήνυμα της ε, διαφάνειας είναι ότι πρέπει να εργαστούμε αμελητή, γρήγορα και να ολοκληρώσουμε ως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου, το αργότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Δεδομένων λοιπόν των περιορισμών που έχουμε στον χρόνο. Για να συνεννοηθούμε λίγο. Χωρίς μικρόφωνο. Ε, θα φύγουμε δικός μετά για τις Βρυξέλλες. Επομένως, μπορούμε να σας διαθέσουμε όσο χρόνο χρειάζεται. Αλλά σε τέτοιου είδου συζητήσει κάποια στιγμή έρχεται και ένα επίπεδο που πια δεν ε, είναι πολύ παραγωγικέ. Αχτουή. Λοιπόν, αυτές τις ε, παρεμβάσεις που έλεγα να τις στα δύο λεπτά, θα τις ορίσω στα τρία. Οι δύο συνεισηγητές πρώτοι. Ιζαμπέλ Τομά, μπορείτε να ξεκινήσετε. Έχετε το λόγο. Καλημέρα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά την Αντιπρόεδρο, όχι μόνο για την παρουσία της εδώ, μας εκθέτει αυτό το ε, έργο, αλλά και διότι πιστεύω πως οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί λάβατε υπόψη μια σειρά από προβλέψεις και ιδέες του Κοινοβουλίου. Και πρώτα απ' όλα την ιδέα ότι πρέπει να τεθεί επιτάπητος πλέον μια αναθεώρηση. Αναθεώρηση που και όσον αφορά βέβαια τις πτυχές της ευελιξίας, παραδείγματι την μην ε, αντιστάθμιση του περιθωρίου για πρόβλεπτες καταστάσεις και γενικά, τα γενικά ε, περιθώρια έχει λάβει αξιέπαινες ε, πρωτοβουλίες και επιλογές, αποδέχεται αυτά τα οποία εμείς είχαμε προτείνει, ιδιαίτερος ε, την δημιουργία ενός ταμείου κατεπηγουσών αναγκών και το διπλασιασμό του ταμείου αυτού. ένα δεύτερο που θα ήθελα να χαιρετήσω από τις προτάσεις σας κάποια επιπλέον ποσά για τις προτεραιότητες της Ένωσης. Χαιρετίζουμε λοιπόν γιατί συμμεριζόμαστε τις προτεραιότητες αυτές. Θα περάσω τώρα σε αυτά που είναι λιγότερο θετικά από τις προτάσεις σας. Ζητώντα συγγνώμη στην αρχή γιατί το έγγραφο δεν το έχουμε λάβει ουσιαστικά ούτε καν επίσημα ακόμα ή πάντω το λάβαμε πριν από πολύ λίγο χρόνο. Δεν μπορέσαμε να το μελετήσουμε στι λεπτομέρειες του. Αλλά υπάρχουν αρκετά προβλήματα που θα ήθελα να επισημάνω. Πρώτον, βλέπουμε τα αριθμητικά στοιχεία για τις δαπάνες, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πόθεν προέρχονται αυτές οι νέε δαπάνες. Έχουμε λοιπόν εν γέννη την ιδέα ότι μπαίνουν στις στα, από τα περιθώρια και πρέπει να δούμε και ποια είναι αυτά τα αποθεματικά γιατί όπως τώρα από τα ανώτατα επίπεδα τα πλαφόν τα έχουμε καλύψει δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλο περιθώριο δηλαδή αλλά θα ήταν καλό να ξέρουμε από ποιους πόρους θα προέλθουν αυτές οι δαπάνες ένα άλλο πρόβλημα αλλά θέστε να μην φαντάζομαι είναι ότι σε σχέση με αυτά τα οποία εμείς είχαμε υπολογίσει επιπλέον ανάγκες ε, απέχουμε πολύ από αυτά τα οποία προτείνετε εσείς Φερρυπίν, εγγύηση για την νεολαία, όπου προτείνεται ένα δις, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια. Εμείς είχαμε πει ένα δις το έτος. Εσείς είπατε ένα δις για τα τέσσερα έτη. Άρα έχουμε πρόβλημα και ως προς τη διάσταση του ζητήματος και πρέπει να το εξετάσουμε. Στις ε, πληρωμές που λέτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εάν δούμε βεβαίως ε, πώς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το έτος νησιν 3 για να λύσουμε το πρόβλημα της αποδέσμευσης των κονδυλίων. Έχουμε ένα πρόβλημα διαφάνειας του προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος Αρτσουή λέει πάντα ότι ο προϋπολογισμός για να είναι καλός πρέπει να είναι ευνόητος για τον πολίτη. Εσείς μας λέτε βέβαια ότι ο πολλαπλασιασμός των ταμείων που είναι έξω από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από τον έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να ζητήματα διαφάνειας, αλλά έρχεστε να μα καταθέσετε αντίστοιχε τέτοιες προτάσεις, περισσότερες, το υπεσοσμό του ΕΦΣΥ, παραδείγματι, του ΕΤΣΕ. Εντάξει, ναι, να τη διπλασιάσουμε την εγγύηση των εγγύσεων, γιατί όχι. Αλλά μετά θα πρέπει να δούμε και πώς θα αξιοποιηθεί το ταμείο αυτό. Μίλησα λοιπόν για την αποδέσμευση των πιστώσεων, μίλησα για το πρόβλημα της διαφάνειας, τα ποσά, την απουσία ένδειξης προέλευσης των κονδυλίων και θα ολοκληρώσω με κάτι πιο γενικό. Η αναθεώρηση μπορεί να καλύπτει πολλά πράγματα, αλλά πάλι μένει μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που εγκρίθηκε το 2013, όπου τα ανώτατα επίπεδα, όπως τα είχαμε εμείς τουλάχιστον ζητήσει, δεν συζητήθηκαν και δεν συζητούνται. Λυπούμε γι' αυτό. Αυτή είναι η πρώτη μου ανάλυση. Λακωνική, ίσως και ασαφής. Αλλά νομίζω ότι αποτελεί, δίνει κάποιες ενδείξεις για το εις κατευθύνσεις που θέλουμε. Ο πρόεδρος. Τώρα το επίπεδο ε, ευελιξίας για τις πληρωμές είπα, είναι βεβαίως ένα άλλο ζήτημα. Παρακαλώ, κύριος Όλμπριχτ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Όταν συζητάμε το ζήτημα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και όταν διαβάζουμε τον κανονισμό του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου βλέπουμε ότι είναι υποχρεωτική μία μετεκλογική αναθεώρηση και ενδιάμεση επανεξέταση του πλαισίου αυτού. Χαιρετίζουμε λοιπόν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει όντω μια πρόταση επανεξέταση και αναθεώρηση. Όντω χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση και δύο τύποι αναθεώρησης προκύπτουν. Θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε απλώς τους πόρους και τις δαπάνες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν κάνουμε μία επανεξέταση των πόρων, δεν έχουμε φρέσκο και νέο χρήμα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε, να ανακατανύμουμε του ήδη φυστάμενου σπόρου στα πλαίσια του προπολογισμού. Η πρόταση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα υφιστάμενα χρήματα. Τι μπορεί επίσης να γίνει με τους ετήσιους προπολογισμούς από το 2017 ω το 2020. Τι θα γίνει με τα επίπεδα πληρωμών σε επίπεδο ετήσιων προπολογισμών και αυτό πρέπει να το δούμε. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόταση αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αν συγκρίνουμε την πρόταση στον, στη δική μας την έκθεση, στο δικό μας το ψήφισμα, το δικό μου και της Ιζαμπέλ με τη δική σας την πρόταση, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία απουσιάζουν. Θεωρούμε πάντως ότι αυτό έχει να κάνει με τη διαφορετική ανάλυση που έχει γίνει. Εμείς αναφερόμαστε όχι μόνο στις υποχρεώσεις αλλά και στα πλεονάσματα που θα πρέπει να προβλέπονται για να έχουμε χρήματα στον προπολογισμό. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο θα αντιδράσει ακόμα πιο βία για το ζήτημα αυτό από ό,τι αντέδρασε για το ζήτημα των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν παρατηθήκαμε και η πρόταση βρίσκεται ακόμα επιτάπητος, ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί, να πρέπει να αντιμετωπιστεί σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο. Με βάση την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να προβλέψουμε και την αντίδραση του Συμβουλίου, να τη φανταστούμε τουλάχιστον. Σίγουρα το Συμβούλιο δεν θα θέλει καμία απολύτω αναθεώρηση. Είναι πάντως σημαντικό να εξηγήσουμε εμείς ότι κάθε φορά που μιλάμε για προπολογισμό που θα βασίζεται σε επιδόσεις και σε αποτελέσματα, προφανώς θα πρέπει να δούμε και την νέα δομή του προπολογισμού, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή κάθε δυνατό μέσο. Πριν από το 2013 υπήρχαν κάποια μέσα τα οποία θα τα χρησιμοποιούσαμε εφόσον αυτό το κρίναμε αναγκαίο. Η στιγμή αυτή έχει έρθει και μάλιστα έχουμε ακόμα μπροστά μας τρία χρόνια πρωτού ολοκληρωθεί το τρέχον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο είναι παρακινδυνευμένη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σίγουρα σύμμαχό σα. Παράλληλα όμω πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο ότι πρόκειται για το πρώτο μόνο βήμα. Γιατί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όχι μόνο για τον απομείναν ίμιση του υφιστάμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Χαιρετήσουμε λοιπόν την πρώτη σε αυτή πρόταση και είναι σημαντικό να δούμε μαζί σας και με το Συμβούλιο το πρόβλημα των πληρωμών. Αναφερθήκατε εσεί στι πιστώσει αναλήψεων υποχρεώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για τι πληρωμέ, για τι πιστώσει πληρωμών. Κεντρικό σημείο τη συζήτηση αυτό και ολοκληρώνουμε το ακόλουθο. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι προτεραιότητες που θέτουμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι την αθεώρηση δεν έχει να κάνει μόνο με χρήματα, έχει να κάνει και με νέες προτεραιότητες. Βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση αναθεώρηση. Πρέπει να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή. Γιατί αν έχουμε προτεραιότητες, ότι θα πρέπει να έχουμε και τα χρήματα για να τις χρηματοδοτήσουμε τις προτεραιότητες αυτές εκτενέστατη συζήτηση έχουμε κάνει με τους βουλευτές στην Επιτροπή αυτή και κάθε φορά βλέπουμε ότι όταν έχουμε προτεραιότητες οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τους απαραίτητους πόρους, τότε χάνουμε απλώς τον καιρό μας. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπετε ότι ήμουν ιδιαίτερα επίοικη με το χρόνο αγόρευση των δύο συνεισηγητών. Από εδώ και πέρα όμω θα ισχύσει πολύ αυστηρό κανόνα των τριών λεπτών. Η κυρία Γκρέσλε είναι η μόνιμη εισηγήτρια για τον δημοσιονομικό κανονισμό και απουσιάζει. Ενδεχομένω ο συντονιστή από το ΕΛΚ θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ναι, θα τα πω πορτογαλικά. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επίτροπο για την πρότασή σας, την πρότασή της και για το γεγονός ότι εμπνευστήκατε στις προτάσεις σας από όσα έκρινε το κοινοβούλιο, ενέκρινε το κοινοβούλιο σε πολύ μεγάλο μέρος, ιδίω το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και με τον όρο αναθεώρηση ε, νομίζω ότι έχουμε πραγματική αναθεώρηση τελικά και θέλω να σας εκφράσω την ικανοποίησή μας. Ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα είναι ικανοποιημένο και το ίδιο και το Κοινοβούλιο. Εδώ μιλάμε για τα προβλήματα των πολιτών και μιλάμε για τόσα θέματα τα οποία αγγίζουν άμεσα τα κράτη-μέλη. Ουδέποτε κατάλαβα την στάση του Συμβουλίου να μην θέλει να ασχοληθεί και να ε, μελετήσει τα είδα τα προβλήματα, να ενσκύψει και να βρει λύσεις. Πρέπει και εκείνοι στο Συμβούλιο να ε, τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών. Μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για απασχόληση. Πρέπει επιτέλου αυτέ οι κοινέ προτεραιότητες τι οποίε όλοι έχουμε συμφωνήσει να γίνουν σεβαστέ. Για το κόσμο, για την έρευνα, για τον ε, μηχανισμό διασύνδεσης τη Ευρώπη, για το Erasmus όλα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν και από τη σκοπιά κυρίως της απασχόλησης και τη απασχόλησης των νέων. 100 ε, ε, εκατομμύρια δεν αρκούν από την πλευρά του, του προπολογισμού και ελπίζαμε ότι το Συμβούλιο θα ακολουθήσει και τη δική μας προτροπή. Πάντως, ε, ε, πρέπει να σας ε, συγχαρώ και για την επιλογή της απλούστευσης που πρέπει να πηγαίνει μαζί χέρι-χέρι με την ευελιξία. Αυτό θέλουμε, να μπορούμε να εκτελέσουμε, να φέρουμε εις πέρα στη Στατική Ευρώπη 2020 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που έχουμε στη διάθεσή μα χωρί να κάνουμε κάποια τεράστια προσπάθεια, δηλαδή να τα ε, χρησιμοποιήσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό τρόπο. Και για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δεν ε, μπορούμε να υπολογίζουμε μόνο με βάση αυτό. Ε, πρέπει να έχουμε και την ανάλογη έγκριση και από το Συμβούλιο. Πρέπει και το Συμβούλιο κάποια στιγμή να αποφασίσει. Πρέπει να βρει μια λύση. Οι πληρωμέ πρέπει να βρίσκονται στο ύψος των ε, δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Αυτό είναι, μια, είναι κάτι το προφανές. Οι δαπάνε είναι άμεσα συνέπεια των δεσμεύσεων. Δεν μπορεί να λέει το Συμβούλιο εντάξει συμφωνώ με αυτό και ε, εγκρίνω και μετά λέει ναι αλλά τελικά δεν θέλω να εκταμιεύσω. Αυτό ε, υπονομεύει την αξιοπιστία μας. Το Συμβούλιο λοιπόν πρέπει να φροντίσει να είναι αξιόπιστο. Πρέπει να φροντίσει και το Συμβούλιο να είναι εξίσου φιλόδοξο όπω το Κοινοβούλιο, γιατί η πρόταση αυτή είναι μεν ευπρόσδεκτη, αλλά εμεί σε πολλού τομεί θα χρειαστεί να την ενισχύσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Γκαρδία Ζαμπάλ, μόνιμη συγγήτρια για τα θέματα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα δημοσιονομικά εργαλεία. Τρία λεπτά. Presidente, en realidad los intervinientes anteriores ya han hecho Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι προλύσαντες νομίζω ότι ανέλησαν πολύ καλά την κατάσταση. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν όντω κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να ξεκινήσω με τα θετικά σημεία. Ουσιαστικά μα λέτε ότι τρει απαιτήσει του Κοινοβουλίου γίνονται σεβαστέ, απλούστευση, μεγαλύτερη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων και ευελιξία. Αυτά είναι τα τρία βασικά αιτήματα που είχαμε υποβάλει εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βλέπουμε ότι όντω έρχεται αποκριθεί στα αιτήματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τούτων λεχθέντων όμω πρέπει να πούμε ότι και η ποσοτικοποίηση 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί μόνο στο 1% από αυτά που έχουμε από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χρήματα αυτά μόνον, αλλά το θεματικό είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τελικά με τα διαθέσιμα αυτά χρήματα. 6,3 δισεκατομμύρια. Από πού θα προέλθουν αυτά δεν είναι σαφέ. Αναφέρεστε σε χρησιμοποίηση περιθωρίων, αναφέρεστε σε υποχρεώσει και δεσμεύσει, αναφέρεστε σε ευελιξία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα το καινούργιο πάντως στην πρόταση αυτή. Δεν υπάρχουν νέοι δηλαδή πόροι, φρέσκο χρήμα και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πιο αρνητικό στοιχείο της πρότασής σας. Μολονότι βλέπουμε κάποιες βελτιώσεις, τελικά η πρότασή σας δεν πηγαίνει πάρα πολύ μακριά. Πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άρα για το 100% του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, πώς θα μπορούσαμε να προβλέψουμε νέους πόρους για τις προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να προωθήσουμε. Ο κύριος Φερνάντες έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι οι ίδιες οι κυβερνήσεις μας κάνουν περικοπές και δεν θέλουν τελικά να απειλήσουν τα ίδια τους τα προβλήματα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις και τα κράτη-μέλη για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω και μία ακόμα επιφύλαξη, μία ανησυχία. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να έχει και ιδίου πόρου. Έχουμε μία ομάδα υψηλού επίπεδου για το ζήτημα αυτό. Θα ολοκληρώσουν σύντομα και την τελική του την έκθεση, αφού το γνωρίζουμε. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ καν στα δικά σα τα έγγραφα, κύριε Επίτροπε, να δούτε καν τον όρο ίδιοι πόροι. Εσείς τι έχετε κατά νου ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των ιδίων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνετε του επόμενου μήνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο σκιώδης εισηγητής, οι σκιώδης εισηγητές μάλλον έχουν το λόγο, Chairman, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Καταρχάς, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου. Εν γέννη, οι προτάσεις σας μας βρίσκουν σύμφωνος, ιδιαίτερα ε, η μεγαλύτερη ευελιξία που θέλετε να εισαγάγετε, την οποία και εγώ επιδιώκω. Το θέμα δεν είναι τόσο πού βρισκόμαστε, αλλά προς τα που κατευθυνόμαστε σε αυτό το ταξίδι, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Βεβαίως, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι επίσης, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και έχω ένα-δύο σημεία να επισημάνω που φαντάζομαι θα μας εξηγήσετε τις λεπτομέρειες. Τρία σημεία λοιπόν που ιδιαίτερως με παραξένεψαν για το ΕΦΣΥ, αξιόλογη επιτυχία του βεβαίως. Τα φιλόδοξα σχέδια για τη συνέχεια όμως ε, μου προκαλούν εντύπωση και οι προτάσει για αύξηση τη χρηματοδότηση. Θα συνεχιστεί όμω από τον τωρινό προπολογισμό αυτή η χρηματοδότηση ή θα είναι νέο χρήμα για να αυξηθεί η προποδότηση του ΕΦΣΥ. Δεύτερο μικρό χρηματοδότηση για τη μετανάστευση τη εγγύηση για την νεολαία. Είναι πάντα βέβαια θέματα που υποστηρίζουμε, αλλά θα ήθελα ναι, επισημάνω ότι πολλές φορές με τις καλύτερες των προθέσεων την ώρα που έρχεται η εκτέλεση, η στιγμή της εκτέλεσης, το κόστος, φέρει πριν για την εγγύηση ε, για την νεολαία, το κόστος άναθεση εργασίας παραγόμενη είναι υπερβολικά υψηλό. Ενώ αυτό που χρειάζεται η νεολαία μας είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία που θα παράγει μόνη τις νέες θέσεις εργασίας. Ας μην ξεχάσουμε λοιπόν και αυτή τη διάσταση. Και κάτι ακόμη, για τις συνεχιζόμενες υποχρεώσεις, αρεξόφυτους λογαριασμούς κτλ. Λαμβάνονται αυτά υπόψη, είναι παρκώς στο πρόγραμμα το οποίο έχετε ε, σχεδιάσει. Θα μπορέσετε να κρατήσετε δηλαδή τον έλεγχο της κατάστασης. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καταρχάς με συγχωρείτε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν άκουσα όλη σας την παρουσίαση. Οπότε αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση, Γιατί έπρεπε να μείνω στην Ολομέλεια. Καταρχάς, να ενώσω τη φωνή μου με αυτή των συναδέλφων που εκφράζουν την ικανοποίησή τους, επειδή αναλάβετε την ευθύνη να προτείνετε όχι μόνο μία review, μια νέα εξέταση, αλλά μία πραγματική αναθεώρηση, μεταρρύθμιση. Αυτό έζητουσε και το Κοινοβούλιο και αυτή ήταν και η στρατηγική που είχαμε συμφωνήσει να θετήσουμε με τους συνεισηγητές. Είναι μια χειρονομία που χαιρετίζω στο σημερινό πλαίσιο με δύο στοιχεία βεβαίω υπόψη. Πρώτον, ότι εξ όσων γνωρίζω τα κάτι μέλη δεν είναι τελείω συνεργάσιμα και να ανοίξουν, ε, τον, να δώσουν τον οβολό τους υπό τις ε, επικρατούσες συνθήκες και έπειτα ότι οποιαδήποτε αλλαγή του πολιτικού του δημοσιονομικού πλαισίου και εδώ κάποιοι το γνωρίζουν πολύ καλά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές και ε, βεβαίως ε, είναι από την αίρεση της ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Αυτό το θυμίζω διότι σε σχέση με κάποια όνειρα που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή κατά νου δεν μπορούμε να κάνουμε δημοσιονομικά όνειρα εάν θέλουμε τουλάχιστον τα όνειρα αυτά να είναι ευχάριστα και όχι εφιάλτες εδώ για το πακέτο που προτείνεται συγκεκριμένα και ιδίω για την απλούστευση που μπορεί να φέρεται με του κανόνε για τι δαπάνε. Να είμαι αρκετά σαφή. Εδώ λέμε απλούστευση. Έτσι. Ε, απλούστευση θέλουμε και να διευκολύνουμε τη δουλειά κάποιων ε, φορεών που αυτή τη στιγμή του έχουν ε, καταβάλει οι γραφειοκρατικοί κανόνε, οι οποίοι είναι απειράριθμοι. Εδώ Κάποιοι από τους ε, κάποιοι από του υπευθύνου τη Επιτροπή μπορεί τελικά να κάνουν ακόμη πιο περιπλοκούς τους κανόνες. Δηλαδή, θέλουμε να δαπάνονται, να δαπάνονται σωστά τα χρήματα και να μην γίνονται πάτες Αλλά όχι κανόνες να τόσο περίπλοκοι που να αποθαρρύνονται οι φορείς και τελικά να ξοδεύουν άδικα την ενεργειά τους. Όχι. Εδώ σε όλε τι ομάδε, και το λέω για όλου του συναδέλφου, και στι μεγαλύτερε ομάδε ακόμα, ότι πραγματικά αυτό που πρέπει να επιτύχουμε είναι η απλούστευση. Ελπίζω ότι υπήρξα σαφή. Επίση ε, και ένα αστιάκι, αν επιτρέπετε, Επίτροπε. Ακόμα και αν δεν είναι ότι καταλληλότερο για αυτή τη συζήτηση, στη σελίδα 6 του γράφου σα βλέπω το εξή λειτουργείται λίγο σαν ε, ένας ε, σύμβουλος του Κοινοβουλίου και ακολουθείται αυτό που θα σας πούμε. Όταν καθορίσατε τον κατάλογο προτεραιοτήτων ε, δεν ζητήθηκε να γίνει ένας συμβιβασμός μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εδώ μιλάμε για έναν ειδικό σύμβουλο της Επιτροπής που ως υπεύθυνο τη Δημοσιονομική Αρχή επίση, πρέπει να παρουσιάσει ένα συνολικό πακέτο και να αποφύγει οποιαδήποτε ε, αμφισβήτηση του πακέτου σε επιμέρους επιτροπές. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας δίνετε αυτή τη στρατηγική συμβουλή ε, και ευχαριστώ για τη συμβουλευτική σας που είναι επιπλέον και δωρεάν. Ευχαριστούμε η κυρία Κυρία Νιριάντα, ευχαριστώ την Επίτροπο ε, Γεωργίευα για τι προσπάθειε που έχει καταβάλει για την πρόταση αυτή. Θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε όλε τι πληροφορίε. Θα συμμεριστώ τι παρατηρήσει των εισηγητών, ιδιαίτερω και των άλλων συναδέλφων. Και εμεί θελήσαμε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών με ομάδε εργασία ε, για τα θέματα αυτά. Η άλλα των προσπαθειών μα. Επίση, στήριξη των πετυχημένων προγραμμάτων και του ΕΦΣΥ, ώστε να αξιοποιούμε καλύτερα διαθέσιμου πόρου και βεβαίω η ευελιξία είναι κάτι το πάντοτε ευπρόσδεκτο. Πρέπει να την εφαρμόσουμε και στην πράξη όμω. Να υπογραμμίσω όπω και οι υπόλοιποι τη μετριοπάθεια στι αυξήσει που προτείνονται ιδίω για, την ε, και την ε, ε, ανάπτυξη. 2,4 δις είναι πολύ παθές ποσό. Πολύ μέτριο. Όπως ε, ανέφερα και προηγουμένως, η απασχόληση των νέων είναι προτεραιότητα και πραγματικά θέλουμε να δούμε ένα δις ετησίως. Αυτή είναι πραγματική επένδυση και συνεχώς μιλάμε για τους νέους. Μιλάμε για την νεολαία σαν να είναι κάτι του μέλλοντος. Όμως είναι κάτι που τώρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι σοβαρό. Και άλλη μία μας μέρημνα είναι ότι προτείνεται την καλύτερη χρήση των δημοσιονομικών εργαλείων. Βεβαίω να ενισχυθεί αυτό ε, ω προ τι ε, ε, αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά να δούμε πώ θα ελεκτρωθούν και ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα. Γιατί πολλοί ε, που χρειάζονται αυτά ω δικαιούχοι είναι οι πιο ευάλωτοι και δεν έχουν πρόσβαση. Θα θυμίσω εδώ τα επικριτικά σχόλια που είχαμε για το πρόγραμμα ΕΦΣΥ και για το γεγονό ότι πραγματικά δεν ωφελεί αυτού που περισσότερο από όλου το χρειάζονται. Και τέλο, κάτι που ανέκαθεν ω Ιρλανδέζα το τονίζω, ο αντίκτυπο του Brexit τι ε, επιπτώσει θα έχει στο εισόδημα και τι επιπτώσει στο σκέλο των δαπανών. Ιδίω για αυτέ τι περιφέρειε και τι χώρε όπω η δική μου που θα πληγούν ε, όλο ιδιαίτερω. Επειδή είμαι από την Ιρλανδία, ε, φανταστείτε μόνο πώ θα μα επηρεάσει, ιδίω για το συνοριακό εμπόριο. Όλα αυτά τα θέματα θα έχουν πραγματικά επιπτώσει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπω το παρελθόν σε να μην έχει γίνει τίποτα. Πρέπει το Brexit να ε, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε στον προπολογισμό, αλλιώ είμαστε χαμένοι πιστεύω. Ευχαριστούμε, κυρία μου. Τώρα ο κύριος Μαραγκάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας, που όντως αποκριθήκατε στην αρχική σας δέσμευση για μια επανεξέταση και αναθεώρηση. Χθες μόνο μπόρεσα να δω το πρώτο σχέδιο του εγγράφου που υποβάλλατε και πραγματικά με γέμισε ελπίδα αυτό. Είδα πολλά θετικά στοιχεία. Πέρα από τα θετικά μου σημεία, πρέπει να δούμε και τα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία μας προσγειώνουν, θα έλεγα λίγο, στην πραγματικότητα. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στην πραγματικότητα. Αν συγκρίνουμε την πρότασή σας με την έκθεση που ενέκρινε η Επιτροπή μας τον Ιούλιο, με την έκθεση δηλαδή Όλμπριχτ Τομά, ουσιαστικά βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μια επικάλυψη στους στόχους μας, υπάρχει μια κάποια σύγκληση Υπάρχει όμως μια απόκληση όσον αφορά το περιεχόμενο, όσον αφορά κάποιες προτάσεις και δυστυχώς η απόκληση αυτή μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η πρόταση τώρα αναθεώρησης είναι κάτι θετικό σίγουρα, αν δούμε όμως πώς έχει πραγματικά η κατάσταση, συνειδητοποιούμε ότι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε είναι εσωτερικές μεταφορές σπόρων ανακατάταξη από τον έναν τομέα στον άλλον. Δεν αλλάζουμε το ίδιο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, επιφέρουμε επιμέρους αλλαγές στο πλαίσιο του MFF. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το πούμε, είναι σημαντικό. Γίνονται κάποιες ανακατατάξεις, ανακατανομές πόρων, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε νέους πόρους πουθενά όσον αφορά την κατάρτιση προτεραιοτήτων. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Συμφωνούμε με πολλά από αυτά τα οποία λέτε, αλλά δεν συμφωνούμε με τις πιστώσεις που προβλέπονται για τα τέσσερα ακόλουθα έτη. Τα όσα λέτε αυτή τη στιγμή για την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων ή τα διάφορα άλλα προγράμματα τα οποία παρατίθεται στην έκθεσή σας. Για κάποια από αυτά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε συμφωνία, για άλλα πάλι όμως δεν συμφωνούμε. Το πιο βασικό ερώτημα είναι το ακόλουθο. Από πού θα προέρθουν όλα αυτά τα χρήματα. Πώ θα χρηματοδοτηθούν όλε αυτέ οι δαπάνε. Αυτό δεν διαφαίνεται καθόλου στο εγγραφό σα δυστυχώ. Τα χρήματα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για την νέα αυτή ανακατανομή πόρων, αλλά από πού θα προέλθουν. Το Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Κρίσεων, το απόθεμα αυτό για την αντιμετώπιση των κρίσεων είναι μια πολύ θετική πρόταση, την οποία χαιρετίζω. Και κάτι ακόμα. Έχω πολλές αμφιβολίες όσον αφορά τις προτεραιότητες που αναφέρεται στον τομέα της μετανάστευσης. Έχουμε την εξωτερική και την εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Διερωτάμε λοιπόν, διατρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε μια εσωτερική αγορά με ασφάλεια και συνεργασία από τη μία πλευρά και από την άλλη να μην έχουμε καταφέρει να διασφαλίσουμε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα τα προγράμματα. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες περιμένουν να εγκριθούν και να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα. Διακόπτει ο Πρόεδρος, ολοκληρώστε παρακαλώ. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να έχουμε μια γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση των κρίσεων που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Κύριε Σάνι, θα αναλάβει ο κύριο Σάνη, παρακαλώ, από το EFTD. Ευχαριστώ πολύ. Επιτροπέ Γεωργίευα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας εδώ σήμερα. Κατά κάποιο τρόπο μετά το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασίλειου αισθάνομαι σαν να βλέπω τα πράγματα απ' έξω από το παράθυρο. Σε ορισμένα πράγματα συμφωνώ απολύτω από τα όσα είπατε ότι πρέπει να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να αποστευθούν οι δομέ, αν και κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια για απλούστευση δομών φαίνεται να υπάρχουν πολιτικά μελήματα και βουλήσει που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Συμφωνώ λοιπόν και πριν από κάνα δύο χρόνια θυμάμαι σας είχα πει ότι κάθε προπολογισμό πρέπει να είναι εστιασμένο και προσανατολισμένο σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και εμένα σε αυτή τη θέση. Ζητήματα όπω επικουρικότητα πιστεύω θα πρέπει ιδιαίτερα να εξεταστούν. Γιατί βέβαια ποιο δεν θέλει τρώγω WiFi, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι σε θέση οι εθνικέ κυβερνήσει να αναλάβουν ε, αυτέ τι ε, πρωτοβουλίε και αποφάσει και θα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι όμως το οποίο δεν γνωρίζουμε τώρα και το οποίο νομίζω ότι ε, διατρέχει όλη αυτή την υπόθεση είναι πότε θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο ίσως, ε, ελπίζω να συμφωνείτε, το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι ξεκάθαρο το ταχύτερο δυνατό ε, το πότε σκοπεύει να θέσει σε λειτουργία το άρθρο 50, ώστε να ξέρουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Brexit. Και δεύτερον, θα ήθελα μια σαφή δήλωση ότι δεν θα υπάρξει από τώρα μέχρι τον Brexit ανατροπή της επιστροφής για τη Βρετανία. Κάτι άλλο. Ποιες είναι οι θέσεις της Επιτροπής σε σχέση με ελληματική χρηματοδότηση σε περίπτωση που το Brexit λάβει χώρα από την ώρα που μιλάμε τώρα μέχρι το τέλος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί είναι χορηγό καθαρό του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένω, μήπω υπάρξει ενίσχυση των προβλημάτων ω προ τι πληρωμέ. Για δε τις περιπτώσεις ε, κάλυψης απρόβλεπτων αναγκών. Έχει ληφθεί κάποια μέρημνα και έχετε διαφορετικά σχέδια ανάλογα με το αν θα φύγει πιο νωρίς από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Βασίλειο ή πιο αργά. Το έχετε καλύψει αυτό, ο πρόεδρος. Ζόλτεκ. Eh δεν είναι εδώ, πολύ καλά. Για να δω ποιοι άλλοι συντονιστές δεν έχουν ακόμη λάβει το λόγο. Κόλμελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ καταρχάς την Αντιπρόεδρο και εγώ για την ε, παρουσίασή της όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, σε πολλά σημεία που αναφέρεται μπορώ και εγώ να συμφωνήσω και να τα υποστηρίξω, Το θεωρώ πολύ σημαντικά. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω πως στο μέλλον θα πρέπει να προσανατολίζουμε τον προπολογισμό μας πολύ περισσότερο σε αποτελέσματα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί να το πει κανείς εύκολα βέβαια, αλλά ε, είναι απαραίτητο να δούμε Όσο πιο δύσκολο είναι στην πράξη να υλοποιηθεί αυτό στα διάφορα κράτη-μέλη. Και έτσι πρέπει να ξανακοιτάξουμε πάνω απ' όλα τους ορισμούς. Πρέπει τα κριτήρια αυτά να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Οι περιγραφές να έχουν κάποια ε, κάποιο απτό αντικατοπτρισμό. Αλλιώ δεν έχει σημασία ό,τι και να κάνουμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα δηλαδή. Να σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λέμε όλοι ότι θέλουμε να ενισχύουμε τι επενδύσει. Βεβαίω, να το δει κανεί έτσι αφηρημένα, πολύ σωστό είναι. Αλλά τι σημαίνει ε, ε, επενδύσει και μάλιστα αιφόρε ή βιώσιμε. Σαν έννοια, σαν ιδέα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βεβαίω μπορεί σε κάθε κράτο να πούμε ότι κάνουμε επένδυση και χτίζουμε χίλιε πισίνε ένα κράτο, Φερρυπίν. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το βιώσιμο ή αηφόρο, γιατί δεν πρόκειται να διατηρηθούν οι, χίλιες, οι, οι αντίστοιχε θέσει για τι χίλιε πισίνε. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε σε όρου πραγματικούς. Δεύτερον, το είπατε και εσείς ότι χρειάζεται διαφάνεια περισσότερη, συμφωνώ και το υπογραμμίζω. Ωστόσο πρέπει να διαρωτηθούμε, είναι όντω υποβοηθητικό της ε, διαφάνειας το να ενισχύουμε τη χρηματοδότηση του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, του ΕΦΣΙ όπου δεν ξέρουμε ακριβώς πώς νέμονται ε, τα κονδύλια κτλ. κτλ. Ή κονδύλια για την Αφρική και είναι στόχοι αυτοί τους οποίους βεβαίως και υποστηρίζουμε και εγώ πολύ συχνά έχω πει στην Επιτροπή μας ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ε, μετανάστευσης, της κρίσης μεταναστευτικής στη ρίζα στο χώρο προέλευσης. Αλλά αυτό δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο με ενίσχυση των κονδύλιων. Χρειάζεται μια σαφής ιδέα για το τι θέλουμε για αυτή την πολιτική και πρέπει να είμαστε σε θέση να περιγράψουμε ποιες είναι οι ακριβώς οι λύσεις που θέλουμε. Δεν μπορεί να είναι μόνο χρήματα, και αυτό το βάζω εισαγωγικά βεβαίω, η λύση. Γιατί θα γίνουμε πιο φτωχοί εμείς, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουν πιο πλούσιοι οι άλλοι στις χώρες αυτές. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σχεδιάσουμε μια πολιτική για τη μετανάστευση, μια πολιτική η οποία θα είναι συνηγμένη στην εθελοντική συμμετοχή. Έχουμε δει ότι συμμετέχουν τα κράτη-μέλη βεβαίως, πρέπει όμως να υπάρχουν και κανόνες ως προς την εθελοντική συμμετοχή για να μπορεί και να προχωρεί ελεγχόμενα η μετανάστευση να είναι πλαισιωμένη με διάφορα μέτρα τα οποία θα αναλαμβάνονται και στις χώρες προελεύσεως. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ε, να μου σχολιάσετε και αυτό το σημείο. Επίσης, σε σχέση με την προοπτική του Brexit, μήπως θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερα και αναλυτικά στοιχεία για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Ευχαριστώ, Τάραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε εδώ πέρα και μας κάνατε αυτή την παρουσίαση και από ό,τι βλέπω ακόμα ονομάζεται το έγγραφό σας αυτό αναθεώρηση Παύλα Επανεξέταση. Άρα θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά τι από τα δύο είναι, έτσι δεν είναι. Και αν θέλουμε πραγματικά να λειτουργούμε πλήρω ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι revision, αναθεώρηση. Αλλά αυτό εξαρτάται βέβαια από τι πολιτικέ ομάδε. Να πω και κάτι ακόμα. Η σημερινή μα συζήτηση με εξέπληξε με τρόπο θετικό, όχι μόνο για αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εκτίμησε όλους ιδιαιτέρως την επικοδομητική προσέγγιση των Alternative for Deutschland και άλλων συντηρητικών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαφόρων ομιλητών από το EFDD. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να εκτιλήσετε η συζήτηση στα πλαίσια ενός κοινοβουλίου, να μπορούν αυτή τη στιγμή να ακούγονται πολλές διαφορετικές απόψεις και βέβαια να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντεμπρέ για την ε, παρέμβασή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα μπορούν να πάρουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δύο λεπτά όμως έχετε ο καθένας. Ολμέιερ παρακαλώ. Ähm, liebe äh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρώτη αυτή επισκόπηση. Τα ερωτήματα τα δικά μου ακολουθούν λίγο πολύ την ίδια λογική και των ερωτημάτων των άλλων ε, συναδέλφων. Έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία ε, ενδείξεις ότι τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να μετακινηθούν προ οποιαδήποτε κατεύθυνση γιατί υπόθηκε βεβαίως με μια κάποια αίσθηση ε, ε, χαριτολογίας ότι χρειάζεται ομοφωνία. Επίσης, το Brexit, τι συνέπειες θα φέρει. Μια-δύο απλές ερωτήσεις διατυπώνω. Η τρίτη. Βλέπω πάντα αυτή την προσπάθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, όπου κέρια σημασία παίρνει η ανάγκη να διαμορφωθεί κατά τρόπο ορθολογικό ένας προγραμματισμός της μετανάστευσης για τα επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχει αποτελέσματα συγκεκριμένα αυτή η βοήθεια. Ερωτώ λοιπόν, τα κράτη-μέλη έχουν κάποια πρόθεση για σοβαρή συνεργασία μεταξύ τους έτσι ώστε να υπάρξει μια σταθεροποίηση στρατηγική αυτών των περιοχών ώστε να μην χρειάζεται να ορίζονται ε, ποσοστώσεις για την προέλευση των ε, ε, μεταναστών οι οποίες κατά πολύ υπολείπονται από τις πραγματικές ανάγκες για την κατάσταση στο Ιράκ που γνωρίζω καλά είναι πολύ χειρότερη από ό,τι νομίζουμε. Στην Αίγυπτο επίσης έχουμε 5 εκατομμύρια πρόσφυγες αυτή τη στιγμή από διάφορες περιοχές. Δεν το έχουμε συζητήσει, δεν τους έχουμε αναφέρει ακόμη, αλλά υπάρχουν στην Αίγυπτο 5 εκατομμύρια πρόσφυγες και αυτό σημαίνει μια σειρά προβλήματα. Και κλείνω λοιπόν Πρόεδρε, ερωτώ, έχετε κάπου διαγνώσει τη βούληση για συνεργασία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Ευχαριστώ Μάνικα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την αισιόδοξη παρουσίαση που μας κάνατε. Ε, βρίσκω θετικό ότι μπορούμε να έχουμε μια θετική στάση εδώ. Ναι, να το μεταφέρετε αυτό και στα κάτι μέλη, να προωθηθεί το ΕΦΣΥ, να δώσουμε μια νέα όθηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στους στόχους μας. Ε, όπως είπατε, και το Κοινοβούλιο συμφωνεί. Εάν θέλουμε να υπάρξει απασχόληση και ανάπτυξη, το growth and jobs τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρξει μια νέα πνοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια όθηση που ε, και με την συνοχή θα πετύχουμε περισσότερη προστατευμένη αξία. Σίγουρα οι προστατευμένοι κανόνε θα μα διευκολύνουν σε αυτό. Και σίγουρα ακόμη ε, οι τράπεζε δυσκολεύονται με τα δημοσιονομικά εργαλεία και με τα χαμηλά επιτόκια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα πνοή, γι' αυτό χρειαζόμαστε την Ένωση των Χρηματαγορών. Δεν αρκεί ε, να παραμείνουμε σε αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για του νέου, χρειαζόμαστε στήριξη στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μας λέτε ότι υπήρξατε πιο συντηρητικοί, πιο επιφυλακτικοί στην προσέγγιση σας, ενώ τώρα βλέπετε ότι το όλο εγχείρημα λειτουργεί, δίνει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό λοιπόν επιτέλους να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα στην πράξη. Η πράξη μας ενδιαφέρει στη χώρα μου, τη Σλοβακία, 86% έχει επιτυχία το πρόγραμμα της ε, απασχόλησης των νέων. Δηλαδή μένουν στην δουλειά τους επειδή έχουν αυτή τη χρηματοδότηση ενώ πριν την χάνανε. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα δεν είχε αξιολογηθεί σωστά ω τώρα. Είχαμε τριμερή συνάντηση το Δεκέμβριο και ο Σλοβάκος ε, υπουργό αναγκάστηκε να αποτιμήσει το όλο πρόγραμμα μέσα σε μία εβδομάδα. Μην χάσουμε πάλι ένα χρόνο γιατί έγιναν όλα αυτά το 2015, το 2016 να προσέξουμε. Και οι ιδέες αυτές να ε, τεθούν σε εφαρμογή ε, άμεσα μέσα σε ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστούμε κύριε Ζούμπιχ. Ναι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την, ε, την Πρόεδρο για την παρουσίαση της πίεση, οι βάρος του ευρωπαϊκού προπολογισμού ενισχύονται ε, και με πιο λίγους ακόμη υπαλλήλου ε, και ως εκ επιβάρος του προπολογισμού έχουμε πολύ μεγάλες ευθύνες να φέρουμε εις πέρα στην εκτέλεση του προπολογισμού. Το θέμα είναι όμως μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι με τόσο στενά περιθώρια. Τα περιθώρια όπου τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τις αποφάσεις, οι τομείς τους οποίους τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τις αποφάσεις αποφάσεις, είναι τα εθνικά ζητήματα και εμείς δεν έχουμε καμία προτεραιότητα. Πώς μπορούμε λοιπόν με όλη αυτή την απλούστευση να διαμορφώσουμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα έχει τους τομείς εκείνους, τους απαραίτητους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα εμπλουτίζει έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε να κάνουμε, να λάβουμε αποφάσεις ε, χωρίς το blending, τη χρηματοδότηση, το σύστημα της σύμπραξης του δημοσιοδοτικού τομέα, ε, ή μάλλον με, την, με τις συμπράξεις, με το blending, με τις χρηματοδότηση, έτσι ώστε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Μουρεσάν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι είναι καλή η πρόταση σε όρους ευελιξίας. Τρία σύντομα ζητήματα. για το αποθεματικό για την κρίση μπορείτε να μας δώσετε τους στόχους ε, πολιτικής που θα καλείτε να εξυπηρετήσει και να χρηματοδοτήσει αυτό το Ταμείο ε, για την κρίση. Ε, πώς θα λειτουργεί, με ποιους όρους θα κρίνετε ότι έχει προκύψει κρίση. Επίσης, τι όγκο χρηματοδότησης προβλέπετε. Γι' αυτό. Δεύτερον, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Υπόθηκε και νωρίτερα και εγώ από την κυρία Τωμά, θυμάμαι καλά, Έχουμε ζητήσει εμείς από το Κοινοβούλιο επίπεδα χρηματοδότησης 1,8 δις ευρώ, επίπεδα δηλαδή χρηματοδότησης ε, των αρχών του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Εσείς τώρα μας προτείνετε ένα δις έως το τέλος του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ο πρόεδρος Γιούνκερ μας είπε το πρωί ότι λειτουργεί ικανοποιητικά και έχει δώσει 9, σε 9 εκατομμύρια νέους τη δυνατότητα εκμάθησης ένταξης σε μια θέση εργασίας. Ερωτώ λοιπόν γιατί να προτείνετε ένα δισεκατομμύριο μέχρι το τέλος του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και έχετε κάποια στοιχεία αξιολόγησης του ε, ταμείου αυτού που θα μπορούσατε να μας δώσετε. Τελευταία παρατήρηση. Η, κάλυψη των ε, κονδυλίων για τον ορίζοντα 2020 και το Connecting Europe βεβαίως είναι πολύ σημαντική, αλλά ε, υπολείπεται κατά πολύ από τα ποσά που είχαν προβλεφθεί πριν από τις περικοπές που έγιναν λόγω του ΕΦΣΥ. Μπορείτε λοιπόν ε, να μας πείτε αν υπάρχει δυνατότητα να ανακτηθούν τα ποσά αυτά, να ανέβουν δηλαδή και πάλι τα ποσά αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Μικρέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και καλώ μιλήσατε για την επικοινωνία. Όντω πρέπει να προβάλλουμε καλύτερα τα θετικά στοιχεία του υπολογισμού, γι' αυτό θέλω να σα ζητήσω και εγώ και να σα ρωτήσω κάτι. Πρώτα απ' όλα το αναφέρατε ήδη. Πολλά δημοσιεύματα είχαμε αυτή την εβδομάδα για το γεγονό ότι πολλά κονδύλια τη πολιτική συνοχή θα αφαιρεθούν και θα κατευθυνθούν στην πολιτική τη μετανάστευση. Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα λένε ότι 25% των κονδυλίων τη συνοχή μπορεί να περικοπούν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λέει τίποτα για το θέμα. Γιατί τηρείται σε και τι θα πείτε όταν επικοινωνήσετε. Διότι πρόσφατα ένα άρθρο έλεγε ότι θα πάρετε χρήματα από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και κάτι θέλουμε να πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Δεύτερο θέμα περί επικοινωνίας ε, το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Στατικό Ταμείο. Θέλουμε το διπλασιασμό του μεγέθου του, ωραίο αυτό, αλλά έχουμε τη στήριξη του κόσμου καταλαβαίνουν οι πολίτε πώ λειτουργεί το Ταμείο, βλέπουν αποτελέσματα, διότι χρειαζόμαστε τη στήριξή του και τη στήριξη των φορολογουμένων για να μπορέσει το Ταμείο αυτό να λειτουργήσει στο μέλλον. Και πάλι λοιπόν αυτά έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Μιλάμε για όλα αυτά τα προγράμματα, όμω ταυτόχρονα το Συμβούλιο μειώνει τη συμβολή στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Είναι, αυτά, είναι αυτές οι δύο ε, συμβατέ. Διότι πολύ ωραία επικοινωνούμε, λέμε ένα σωρό πράγματα ότι θα κάνουμε, αλλά τα κάτι μέλη τελικά δεν συμφωνούν. Και ε, επιτά μιλήσατε για την ε, ε, απασχόληση των νέων και το σχετικό πρόγραμμα. Είναι πολύ καλό πρόγραμμα, πολύ καλή πρωτοβουλία. Επίση είπατε και για το Wi-Fi for you. Είναι πολύ καλέ όλε οι ψηφιακέ πρωτοβουλίε. Απλώ να πω ότι ω επαγγελματία βλέπω ότι θα αργήσει να πραγματοποιήσετε αυτό σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την επικράτεια, αλλά αναφέρατε ένα ποσό 15 εκατομμύρια ευρώ. Ε, αρκεί αυτό για να υπάρξει Wi-Fi ελεύθερο και δωρεάν ε, σε όλη την Ευρώπη. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριο Τενανού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να πω στον συνάδελφο Ντεπρέ ότι δημοσιονομικά νο, όνειρα μπορούμε να κάνουμε συνέχεια. Εγώ ονειρεύομαι νύχτα και μέρα τέτοια πράγματα. Και τι ονειρεύομαι, το κοινοβούλιο να έχει εδώ το λέγειν του και να εισακουστεί. Και να έχει και ίδιου πόρου που να το επιτρέπουν, επιτρέπουν όντω να αναλάβει δράση. Διότι εάν έχουμε πόρου από τον οποίο να μπορούμε να οργανώσουμε τη δράση μα, ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλιώ τελικά πρέπει να στραφούμε σε δημοσιονομικά εργαλεία που δεν εξασφαλίζουν καμία καλή συνέχεια για το μέλλον. Όπω το πρόγραμμα Juncker. Πολύ ωραία ιδέα ήταν, αλλά η χρηματοδότηση είναι το πρόβλημα και η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι κάτι που θα εγγυηθεί σε ένα δημιούργημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσει. Αυτέ οι πρακτικέ λοιπόν κάπω με ανησυχούν, όπω και με ανησυχεί το αν θα υπάρξει ένα ταμείο για την Αφρική. Από όσα γνωρίζω για την Αφρική και την γνωρίζω καλά, μπορώ να σα πω ότι όταν επισκέφτηκα την ε, περιοχή με την οποία συνεργαζόμαστε στην Αφρική, με πήγα να επισκεφτώ ένα κέντρο που παράγει συγχρονότατο εξοπλισμό και εκεί ε, υπεύθυνοι, που, υπεύθυνοι που είχαν αναλάβει ήταν ε, Κινέζοι. Αυτοί παρήχαν ε, όλη τη διοικητική, οργανωτική και ε, εμπειρογνωμοσύνη. Ε, εκεί απουσιάζουμε πλήρω. Η Αφρική είναι μια ήπειρο με πολύ μεγάλο δυναμικό. Η Ευρώπη λοιπόν θα έπρεπε και θα όφιλε να είναι πολύ περισσότερο παρούσα στην Αφρική. Όχι μόνο να αφήνουμε την πρωτοβουλία στου ιδιώτε και στι ιδιωτικέ επιχειρήσει, αλλά να υπάρξει μια πραγματική βοήθεια προ την ανάπτυξη τη Αφρική. Αυτό είναι σημαντικό να ακουστεί ξανά και νομίζω ότι επί του θέματο θα έπρεπε και θα ήταν προ τιμήν τη Επιτροπή και του Κοινοβουλίου και όλων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων να κάνουν κάτι προ αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μιλάμε για μια πολιτική που προχωράει με μικρά βήματα. Εγώ ε, συγχαίρω την Αντιπρόεδρο που προχώρησε λίγο στα θέματα αυτά. Είναι πολύ λίγα αυτά που έγιναν, αλλά είναι ήδη κάτι. Το θέμα είναι λοιπόν να κοιτάξουμε να κάνουμε όνειρα ακόμη πιο πέρα και για το απότερο μέλλον. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου. Ξέρετε, τι διακρίνει την Κίνα τις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η Κίνα έχει έναν κεντρικό προπολογισμό, ε, ένα δημόσιο προπολογισμό, ενώ η Ευρώπη έχει κρατικά χρέη. Ε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω τσεχικά, θα είναι καλύτερα. Δεν Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Αντιπρόεδρε, Θυμάμαι την ακρόασή σα, ήταν εξαιρετική. Ήταν από τι καλύτερε ακροάσει που έλαβαν χώρα εδώ. Ε, και το είπα και σε όλου του δημοσιογράφου. Ε, είχατε πει τότε κάτι καθοριστικό, το οποίο ήταν φοβερά ενδιαφέρον και πηγή για μένα. Μα είπατε τότε ότι θα κοιτάξετε να υπάρξουν ήδη οι για τη χρηματοδότηση. Αυτό Πραγματικά το είχα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη και θα σας στηρίξω όπως σας στήριξα και τότε. Θα σας στηρίζω και στο μέλλον. Σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτή τη διερεύνηση, πόσο μακριά έχετε πάει. Υπάρχει μέλλον. Η Ευρώπη βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση από το παρελθόν. Αυτό είναι σαφές. Όμω, μα είπατε, ε, και το είχατε πει μάλλον στο παρελθόν, και ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα πάμε ακόμη μακρύτερα. Αλλά ναι, ναι θέλω να δω πρωτοβουλίε ε, όπω αυτή για του νέου να συνεχίζονται. Καλά κάνουμε και τα συζητάμε. Προφανώ, εγώ πιστεύω ότι οι νέοι θα βρουν την άκρη του. Εγώ χάσα τον πατέρα μου όταν ήμουν 18, αλλά κατάφερα να ιδρύσω τρεις πολύ επιτυχημένε μικρέ εταιρείε. Οι συνάδελφοι ανέφεραν κάτι που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήταν διακριτική μεταχείριση οι Νορβηγοί να, να πληρώνουν 144 144 ε, λίρες ε, κατά κεφαλή και οι Έλληνες μόνο 64 ε, στη συνεισφορά του στον προπολογισμό. Μήπως αυτό πρέπει να το ε, αλλάξουμε, μήπως πρέπει να δούμε ποιος πληρώνει τι ξανά. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου που είναι γεμάτες πρόκληση. Ευχαριστούμε. Εάν το Brexit ε, μας χρησιμεύσει για να ευθυγραμμιστούμε την Νορβηγία, ίσως καλύτερα. Η κυρία Μπάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε για, τις, ε, για την παρουσία σας. Έχω ερωτήσει σε δύο θέματα. Το ΕΦΣΥ, καταρχάς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ξέρετε ότι οι πράσινοι έχουν επικριτικά στα θέματα του ΕΤΣΕ, ιδιαίτερα ως προς ε, την απουσία για τις περιφέρειες της επενδύσεις. Δηλαδή δεν στοχεύονται ιδιαίτερα οι περιφέρειες με υψηλά επίπεδα ανεργίας ή άλλες αντίστοιχες ανάγκες. Και η δεύτερη ερώτηση για την ε, παράταση και την αύξηση των ποσών. Παράταση διάρκειας και αύξηση των ποσών. Έχει ζητηθεί αυτό ε, για το έτσε υπάρχουν δηλαδή ποσοστός όπως προβλέπατε και στην περιφερειακή πολιτική για τις επενδύσεις στην κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές επενδύσεις όπως είπα προβλέπονται αυτά ήδη στην πολιτική της συνοχής εδώ και καιρό. Και δεύτερη ερώτηση για το gender budgeting ε, για την ενσωμάτωση δηλαδή, της τάσης του φύλου εν γέννη ε, στην πολιτική και προγωγή της ισότητας του διαφορού τομείς. Είναι θέμα δικό σας το ξέρω. Στην τελευταία δημοσιονομική περίοδο στο πλαίσιο του του δημοσιονομικού πλαισίου είχαν ε, διατυπωθεί αρκετέ εκθέσεις, είχαν καταρτιστεί αρκετέ εκθέσει για το βαθμό στον οποίο ο ευρωπαϊκό προπολογισμό μπορεί να ωφελεί την ισότιμη μεταχείριση και στι ευκαιρίε για άνδρε και γυναίκε. Έχετε λάβει και αυτή τη διάσταση υπόψη στο προσοχή προπολογισμό. Ευχαριστώ, Νόβακοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω και εγώ να μιλώ για δημοσιονομικά όνειρα όπως και εσείς. Ίσως κάποιο νερό μου δημοσιονομικό να υλοποιηθεί. Το Horizon 2020, το Erasmus Plus. Θα πρέπει να πω τώρα προσοχή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε με του νέου και να του πούμε ότι θέλουμε να του βοηθήσουμε, θέλουμε την καινοτομία, αλλά κόβουμε κατά 8% τα κονδύλια, ή ότι είμαστε ενδιαφέρουν πολύ οι νέοι και θέλουμε να του βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ούτε καν τα μισά από τα προγράμματα που κατατίθενται στο πλαίσιο του Erasmus Ξέρω ότι η κρίση βεβαίως την οποία διανύουμε είναι μια κρίση σκληρή. Θα τελειώσει όμως. Μπορεί να μην τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα τελειώσει κάποια στιγμή. Και θα ήθελα να μην εγκαταλείψουμε τις προτεραιότητές μας στην περιγραφή ε, του αύριο για, για τη στιγμή που θα έχει τελειώσει αυτή η κρίση. Διαφορετικά θα έχουμε, δώσει, θα έχουμε μετακυλήσει τις προτεραιότητές μας σε άλλους τομείς. Επίσης, ε, οι καθυστερήσεις που είχατε ως προτεραιότητα ορίσει από πέρσι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, η πρόταση για τη μείωση πληρωμών σε σχέση με την πολιτική συνοχής 3,9% και αύξηση των πληρωμών για τη μετανάστευση με 24,2%. Πώς θα επηρεάσει τις καθυστερήσεις πληρωμές. Οι καθυστερήσεις πληρωμές είναι κάτι σαν την παχυσερκία στο υπροπολογισμό. Όσο συνεχίζουμε να ε, μην εκτελούμε λογαριασμούς, να μην ε, εξοφλούμε λογαριασμούς, όλο και διονγκώνεται αυτή η καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Σαρβαμά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου πολύ σύντομα να πάρω το λόγο μετά από τους συναδέλφους να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Πρώτον, όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και πώς έχει πραγματικότητα το τρέχον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το μέγιστο που μπορεί να γίνει. Τελεία και παύλα. Όλοι θα θέλαμε περισσότερους πόρους, όλοι θα θέλαμε κάτι παραπάνω. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι ότι ε, έχουμε τουλάχιστον μία αναθεώρηση η οποία μπορεί να αποτελέσει και επανεξέταση και αυτό αποτελεί τώρα πραγματικότητα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο μέλλον. Γιατί έχει τελειώσει ο διαθέσιμος χρόνος και είναι οι πρωτεύουσε στα κράτη-μέλη που τελικά θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις δηλαδή, ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς κάνουμε κάθε τι το δυνατό στα πλαίσια της δικής μας Επιτροπής, ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους και τους λέμε κοιτάξτε πρέπει να εργήσετε με αυτόν τον τρόπο, αλλά η τελική ευθύνη βαρύνει τις κυβερνήσεις. Αναφέρομαι τώρα στην περίοδο μετά το 2020. Σχεδόν έχουμε φτάσει το 2017. Αν είμαστε λοιπόν πραγματικά ειλικρινεί, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι η περίοδος μετά το 2020 θα είναι η πλέον καθοριστική περίοδος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται ανακρι... ολοσχερής επανάσταση στα πλαίσια του προπολογισμού, αλλά οι βασικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από τις ίδιες κυβερνήσεις. Ελπίζω ότι εσείς μπορείτε να στείλετε αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνταχθούν στον αγώνα αυτόν. Πρόεδρος, δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω κάποια πράγματα, αν μου το επιτρέπει η Επίτροπος. Καταρχάς, χαιρετίζω πραγματικά την όλη ευφυΐα που διέπει αυτή την πρόταση. Αν κατάλαβα καλά, τα ανώτατα όρια δεν τροποποιούνται. Ωστόσο υπήρχαν κάποια περιθώρια τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, επομένως εσείς προτείνετε αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε δημοσιονομική πρακτική, υιοθετώντα μεγαλύτερη ευελιξία και προσπαθώντας παράλληλα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που είχε προκύψει ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις δύο αρμόδιες για τον προπολογισμό αρχές δηλαδή, το γεγονός ότι ε, τα μέσα ευελιξίας μπορούσαν να ανεπερβούν τα ανώτατα όρια όσον αφορά τις υποχρεώσεις, αλλά όχι για τις πληρωμές. Στα πλαίσια λοιπόν της συνοθεώρησης αυτής θα μπορούσαμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό και να δικαιώσουμε τελικά και αυτό που είχε πει τότε το Κοινοβούλιο, ότι μπορούμε να υπερβούμε δηλαδή τα νότατα όρια και για τις υποχρεώσεις και για τις πληρωμές. Και βέβαια θα πρέπει να προχωρήσουμε και με την απλούστευση την οποία αναφάρεται. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν προβάλλουμε προς τα έξω την καλύτερη δυνατή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν ορισμένοι φορείς οι οποίοι δεν ζητούν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί πολύ πολύπλοκα. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των προτέρων θέλει να κρίνει για συγκεκριμένα προγράμματα, για θα πρέπει να εγκριθούν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ο έλεγχος να γίνεται εκ των υστέρων. Είδαμε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί, δεν έχουν εγκριθεί, ενδεχομένως επειδή είναι αρκετά πολύπλοκες, αλλά και επειδή ορισμένοι φορείς από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καλύπτουν 100% τις δαπάνες και υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε πολύ δεινή κατάσταση γιατί αν αποδεχθούν τα κοινοτικά κονδύλια αυτό συνεπάγεται το ότι θα πρέπει να χρεωθούν και τα ίδια στη συνέχεια, να συμβάλλουν μέσω δικών του δημόσιων δαπανών. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν Αντί να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια συνοχής, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο άλλους τομείς, άλλα προγράμματα, όπως τον ορίζοντα 2020, προκειμένου να αποφεληθούν τα κράτη-μέλη για κρατικά προγράμματα, χωρίς να περνούν απαραίτητα από τα κονδύλια συνοχής. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι οι αποδεσμεύσεις πιστώσεων και η κατάργηση προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις μελλοντικέ δαπάνες που πρέπει να γίνουν υπέρ των κρατών χωρίς να χρεωθούν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ολοκληρώντα λέγοντα ότι το όνειρο πρέπει να συνεχιστεί, το είπε κάποιο επίση ότι ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια διεξοδική ανάλυση λοιπόν τη πρότασή σα. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Thank you very much for the... Uh, Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις και τη γενική θετική σας τάση. Ε, να είστε βέβαιοι ότι έχουμε στρέψει το βλέμμα πολύ ψηλά στον ουρανό. Αλλά τα πόδια μας πατάνε γερά και στη γη και στην πραγματικότητα. Ζητώ συγγνώμη που δεν ξεκίνησα ευθύς εξ αρχής με δύο πολύ απλές διευκρινήσεις. Πρώτον, σεβασμός για τα άνωτα όρια, η πρόταση αναθεώρησής μας είναι μέσα στα όσα ορίζονται από τις τεχνικές παραμέτρους για τις οροφές, τα όνοτα τα όρια. Και δεύτερον, θα επανέλθω σε αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει όθηση για να γίνουν περισσότερα περί ειδικών εργαλείων, θα θέλαμε να λύσουμε προβλήματα που σέρνονται εδώ και πολύ καιρό. Και μετά, από πού ε, ήρθε, από πώς μας ήρθε αυτή η αναθεώρηση. Επειδή έχουμε περιθώρια από τα κεφάλαια 2 και 5, που ήταν η βασική πηγή και τα οποία ήταν τα μη δεσμευμένα ποσά είναι αυτό φρέσκο χρήμα ή όχι. Ε, όχι, είναι εντό του χαρτοφυλακίου δεσμεύσεων που έχουν οριστεί από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμω είναι χρήμα που από την άποψη των ε, προγραμμάτων που θα επωφεληθούν είναι φρέσκο χρήμα, είναι νέοι ε, επιπρόσθετοι πόροι. Τώρα, έχω να κάνω μια σοβαρή ειδοποίηση για την πραγματική ε, προσθετικότητα, σωρευτικότητα μάλλον. Πρώτον, εάν το Συμβούλιο συμφωνήσει στη δημιουργία ενός ταμείου αντιμετώπισης των κατεπηγόντων από τα ποσά τα οποία δεν έχουν δεσμευτεί, αυτό είναι πρόσθετο στα όσα έχουμε προβλέψει, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επαφιόμαστε στην ε, πρώτερη δημοσιονομική μας άσκηση. Δεύτερον, εάν το Συμβούλιο συμφωνήσει στο διπλασιασμό του εργαλείου ευελιξίας και της αντιμετώπισης κατευθυγόντων, αυτό θα μας δώσει 750 εκατομμύρια που δεν θα τα είχαμε ιδάλλως. η πιο σημαντική, όχι δέσμευση, αλλά πληρωμή, ο παράγοντας πληρωμής δηλαδή, θα υπάρξει εφόσον γεφυρωθεί η διαφορά απόψεων κάποιων κρατών στο Συμβούλιο, όχι όλων, μερικών κρατών στο Συμβούλιο και Επιτροπής και Κοινοβουλίου για το αν οι πληρωμές για τα ειδικά εργαλεία είναι πρέπει να τεθούν πάνω ή κάτω από τις οροφές. Όπως ξέρετε, ως τώρα δεν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε στο σημείο αυτό και βασιστήκαμε στο γεγονός ότι υπάρχει χρόνος για να επιληθεί Και αυτό που κάνουμε συνήθως ε, στην Ευρώπη όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα, δηλαδή να κλωτσάμε τον τενεκέ ε, στο χωράφι μέχρι να μην το βλέπουμε άλλο. Δεν θα υπάρχει εδώ όμω ο τενεκέ το, πια, το τενεκεδένιο κουτάκι για να το κλωτσίσουμε. Δεν θα υπάρχει ούτε το χωράφι πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε ε, και να βάλουμε τις πληρωμές πάνω από τις οροφές με την πολύ απλή δημοσιονομική συλλογιστική, ότι οι πληρωμές ακολουθούν τις δεσμεύσεις. Εάν οι συμπεφωνημένες μας δεσμεύσεις είναι πάνω από τις οροφές, είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε ότι οι πληρωμές θα είναι κάτω από τις οροφές. Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα αυτό, είναι εντελώ πολιτικό και γι' αυτό ε, πρέπει να συζητηθεί μαζί με τα άλλα πολιτικά σημεία της συζήτησης. Ρώτησα ποιο είναι το αίσθημα που επικρατεί στο Συμβούλιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι δύσκολο να το φανταστείτε. Το Συμβούλιο τίνει να προτιμά να υπάρξει review και όχι revision, δηλαδή να αναθεώρηση, απλώ ενδιάμεση αποτίμηση. Στην επίσκεψή μου στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ, όλοι οι υπουργοί και όχι μόνο όσοι ε, έχουν ιδιαίτερες απόψεις ε, έδειξαν ε, σχετικό, σχετικά περιορισμένο ενθουσιασμό για το σύνολο του πακέτου. Τώρα, έπρεπε να επιλέξουμε κάτι που να είναι ήπια αναθεώρηση. Δηλαδή, τα προγραφτικά όρια που έδειξε το Συμβούλιο μην ξεπερνάτε τις οροφές. Αντικειμενικώς υπάρχει περιθώριο για συζήτηση και θα φροντίσουμε να προβάλλουμε τα επιχειρήματά μας βασιζόμενοι στις συζητήσεις που έχουμε με το Συμβούλιο και ε, ακόμη πιο σημαντικά για το πολύ σημαντικό γεγονός ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την σώρευση προτεραιοτήτων χωρίς τους ανάλογους πόρους ε, για αυτές. Οι προτεραιότητες αυτές πολύ συχνά ε, έρχονται από το ίδιο το Συμβούλιο. Αυτό που θα καθορίσει την επιτυχία την αποτυχία μας, για να είμαι εντελώ ε, ομοί, είναι πόσο θα καταφέρουμε να πείσουμε το Συμβούλιο ότι η δέσμευση να είμαστε σταθεροί στις προτεραιότητες, ακόμα και αν είναι αρνητικές, εάν αυτή η δέσμευση ισχύει. Και αν οι δεσμεύσεις μας να βρούμε λύσεις θα υπερισχύσουν. Έχουμε ανέκαθεν φανεί αποτελεσματική στο να αναλάβουμε νέες προκλήσεις ε, και νέες προτεραιότητες που χρειάζονται αντιμετώπιση. Στη γραμμή στον προπολογισμό υπάρχει ε, ειδική ε, γραμμή, πόρτα εξόδου για τις νέες προτεραιότητες αλλά και για τις παλιές. Πρέπει να δείξουμε λοιπόν πυγμή ώστε να χτίσουμε ένα σπίτι που να στέκεται καλύτερα στα πόδια του. Διότι αυτό αφορά την καρδιά της αξιοπιστίας μας. Και με τα δύο σκέλη της δημοσιονομικής αρχής να ισορροπούν. Βεβαίως, είναι σαφές για μένα. Έχουμε πολλή δουλειά όλοι μας για την αξιοπιστία του σκέλους των δαπανών του προπολογισμού. Έχουμε επιτελέσει θετική πρόοδο τώρα και πρέπει να συνεχίσουμε αμήλικτοι, διότι μόνο αν φανούμε αμήλικτοι, τότε μπορεί να καταφέρουμε να ξαναδούμε με ένα βλέμμα προς την αύξηση και τους ίδιους πόρους τα εισοδήματα, το κομμάτι των εισοδημάτων του προπολογισμού. Αυτό έχει τεθεί πολλές φορές στο ανώτατο, στην ομάδα ανώτερου επίπεδου ε, τα θέματα αυτά των εισοδημάτων του προπολογισμού, των πόρων του προπολογισμού. Ε, συμμετέχω και εγώ ίδια και η Επίτροπη Μοσχοβησή και Τίμερμανς και για την ώρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αυξήσουμε τις πηγές έβρεσης ίδιων πορών εκτός και αν αποδείξουμε ότι είμαστε καταπληκτικοί στο πώς κάνουμε τις δαπάνες στο σκέλος των δαπανών του προπολογισμού. Δεν υπάρχει καμία ε, περίπτωση για ελαφρά την καρδία χρήση χρήματος, εκτέλεση ποσών και η επιφυλακή του Συμβουλίου είναι τεταμένη ιδίω, τεταμένη μάλλον ιδίως ως προς την λογοδοσία στους πολίτες. Πρέπει το περιθώριο λιγμό που έχουμε να ευθυγραμμιστεί με τις βασικές μας προτεραιότητες. Και θα ξεκινήσω με κάτι που ανέκυψε πολλές φορές στην κουβέντα, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Εκτιμώ το επιχείρημα πολλών ότι ένα δις ετησίως είναι αυτό που πραγματικά θα εξασφάλιζε τη συνέχεια. Έχουμε δύο δις, όχι ένα στην πραγματικότητα. Ένα από αυτό το πακέτο και ένα από το κοινωνικό ταμείο. Και θέλω να το τονίσω και πάλι. Εάν η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ε, ανεργίας των νέων. Υπάρχουν 4,6 δις ευρώ στη διάθεσή του που είναι προορισμένα κυρίω για εκείνε. Εάν λοιπόν λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην έχουμε ένα ετησίως, εάν ανασκουμποθούμε. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πληρωμές πάνω από τα ανώτατα όρια, δεν μπορούμε, αλλά για καθένα από τα λύματα του προπολογισμού που σα παρουσίασα μπορεί και έχει κάθε λόγο να εγκριθεί. Εγώ και οι συνάδελφοι μου στο Σώμα των Επιτρόπων ε, στηρίζουμε την πρόταση κυρίω γιατί αισθανόμαστε ότι είναι δίκαιοι δεν υπάρχει καμία ε, συνεννόηση κάτω από το τραπέζι, ε, στα παρασκήνια, αλλά κοιτάμε να κάνουμε δίκαιες και αποτελεσματικές προτάσεις. Νομίζω και γι' αυτό πιστεύουμε ότι τα 4,6 δις πρέπει να είναι μέρος ε, της συζήτησης, όταν θα δούμε το πού θα πηγαίνουν τα χρήματα, διότι υπάρχουν και τα άλλα προγράμματα. Ναι, θέλουμε να αποκαταστήσουμε ποσά στον προπολογισμό κονδύλια τα οποία περικόψαμε πριν για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το έψη. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με την πρότασή μας αυτή για να στηρίξουμε αυτά τα προγράμματα. Δυστυχώς μας έπληξε αυτή η μείζον μεταναστευτική κρίση και άσκησε πιέσει στον προπολογισμό που προ... προηγουμένως δεν υπήρχαν. Πρέπει λοιπόν όλοι να κοιτάξουμε με προσοχή τα προβλήματα που τίθενται ενώπιόν μας και να φανούμε όσο το δυνατόν πιο μετρημένοι και ζυγιασμένοι στις αποφάσεις μας μπορούμε. Θέλουμε να κάνουμε και κάτι ε, που μας το ζητάει και το Κοινοβούλιο. Τα δημοσιονομικά εργαλεία στην ε, ε, διευκόλυνση και σύνδεση της Ευρώπης δεν λειτουργούν πολύ καλά. Παίρνουμε κάποια ποσά για να στρίξουμε το δεύτερο εύση, κάποια μόνο, αλλά θα τα δώσουμε σε δωρεές. Δηλαδή, και πάλι, στο πνεύμα της ισόρροπης, ορθολογιστικής, ζυγισμένης προσέγγισης που ακολουθήσουμε, να καθορίσουμε τα σωστά βήματα, ένα προς ένα, όπως τα περιέγραψα. Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή, αυτό το απόθεμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, αυτό το ταμείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, με τι χρήμα, τι ποσό, από πού και για πόσο. Έχουμε το προηγούμενο του παρελθόντος, 3 ως 4 δις ευρώ αυτό θα είναι το ποσό, αυτό θα είναι η οροφή, το εργοτόριο και μετά θα δούμε πού μεταξύ του 3 και του 0 μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ως προς το τι θα κάνει, τι θα επιδιώκει. Θα καθορίσουμε δείκτες κρίσης, διότι δεν θέλω να λέμε μόνο για τέτοιου είδους κρίσεις τα εκταμιεύει. Αυτό που είδαμε τα τελευταία 7-8 χρόνια είναι ότι η κρίση έρχεται με αρκετά γενή τρόπο. Δεν την αναγγέλει κανείς ε, στις πύλες, ε, ούτε προειδοποιεί για την άφηξή της. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα μαξιλαράκι για την επόμενη κρίση. Δεν ξέρω ποια θα είναι, δεν ξέρω από πού θα έρθει, αλλά θα έρθει και θα μας πλήξει. Ε, και πρέπει, όπω βλέπουμε την τωρινή κρίση, να υπάρχει ήδη ένα μηχανισμό λογοδοσία. Αυτό μα ενδιαφέρει. Μα ρωτήσαν τι θα κάνουμε και ποια είναι η στατική μα για του μετανάστε και τι πρόσφυγε. Ξέρετε, το είπα και προηγουμένω. Εδώ στην Ευρώπη πρέπει να είμαστε πιο περήφανοι για το πώ το χειριστήκαμε αυτό το θέμα. Ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλου. Δεν ξέρω καμία χώρα η περιφέρεια του κόσμου που 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι θα έφταναν σε ένα χρόνο και αυτό δεν θα δημιουργούσε τεράστιο σοκ. Όμως ε, σταδιακά και κάποιες φορές και με σφάλματα, αλλά αντλώντας και διδάγματα από αυτά, έχουμε δημιουργήσει μια πιο νερομονισμένη κοινωνική προστασία. Οι χώρες δεν είναι εντελώ απροετοίμαστε, ούτε τόσο μακριά μια από την άλλη. Έχουμε αναγνωρίσει τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, ώστε να γνωρίζουμε ποιο έρχεται και το είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ δεν μπορούμε να ε, φορέσουμε με το ζόρι σε όλους τον ίδιο κορσέ. Ε, πρέπει να φροντίσουμε με τους μετανάστες να αποδεχτούμε και τις διαφορές μας και να έχουμε μια νέα αντιμετώπιση με τις διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις μας. Εάν δούμε λοιπόν και αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να γίνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε τα γενεσιουργά αίτια, θα καταλάβουμε ότι εάν οι πρόσφυγες λόγω χάρη δεν μπορούν να εργαστούν στην Ιορδανία, δεν πρόκειται να μείνουν στην Ιορδανία, Εάν όμως δημιουργήσουμε μία διευκόλυνση εμπορίου που να επιτρέπει στις εταιρείε τα προϊόντα των προσφύγων να φτάνουν στην αγορά μας, τότε η Ορδανία μπορεί να αλλάξει και τη στάση της, όπως ήδη κάνει. Άρα είναι πολλά αυτά που μπορούμε να διδαχθούμε από την κρίση και να προσαρμοστούμε σε αυτά που θεωρούμε τώρα μια ε, απόκριση συστηματικά και ενοιολογικά καλύτερα δομημένη. Γι' αυτό έχω την αυτοπεποίθηση να λέω ότι 3,9 δις πρέπει να πάνε εκεί. Υπάρχει και μια πολύ σημαντική παρατήρηση για το συσχετισμό μεταξύ επενδύσεων και ε, θέσεων εργασία. Με άλλα λόγια, το ΕΦΣΥ δεν αφορά μόνο τις επενδύσεις, αφορά και τις θέσεις εργασίας. Ίσως είναι καλύτερα για τους νέους ο, ειδικός, ο ιδιωτικός τομέας να δημιουργήσει ευκαιρίες και πρωτοβουλίες για αυτούς, παρά να προσπαθήσουμε εμείς μέσα από τον δημόσιο τομέα να δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα, ε, προσπαθώντας να φτιάξουμε θέσεις εργασίας. Πρέπει να αναζητήσουμε όλους τους δυνατούς τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Ευρώπης. Νομίζω αυτός είναι ο τρόπος που θα πρέπει να προχωρήσουμε. Μας ενδιαφέρει να είμαστε καλύτερα διασυνδεδεμένοι. Όχι να είμαστε απομονωμένοι, μονωμένοι ο καθένα στη γωνιά του. Και δέχομαι και την παρατήρηση για την ε, προτίμηση, για την επιλογή του Wi-Fi for you και αν αυτό είναι πραγματικά δυνατό να το καταφέρουμε με δημόσιο χρήμα και μόνο. Το συζητήσαμε με του υπευθύνου του προπολογισμού, ειδικά αυτό το ζήτημα, και καταλήξαμε στο συμπεράσμα ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εναρμονιστεί η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην καλύτερη πρόσβαση όλων, όλων των πολιτών. Οπότε η Εστονία δεν θα είναι ένα βασίλειο WiFi σαν νησίδα και η πέθρο τη Βουλγαρία θα είναι κατά 60-70% χωρίς καμία ψηφιακή δυνατότητα. Ε, μπορεί να σας ακούστε και έτσι όταν μίλησε ο Πρόεδρος, αλλά αυτό που λέμε δεν είναι δωρεάν πρόσβαση για όλους. Δεν είναι αρχή της αγοράς αυτής, αυτός, αυτή δεν είναι ο σωστός τρόπος. Αυτό που προτείνουμε είναι ένα πρόγραμμα 50 εκατομμύρια συν 70 που ήδη υπάρχουν για να δημιουργηθεί ένα σύστημα δελτίων το οποίο θα επιταχύνει τη δυνατότητα οι δημόσιοι χώροι να γίνουν hub καινοτομίας και πρωτοπορίας, να γίνουν πραγματικά κέντρα γι' αυτό. Ναι, με τα voucher πιστεύω ότι θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Δεν είμαι βεβαίω εμπειρογνώμων, αλλά αν έχετε ιδιαίτερε παρατηρήσει ε, είναι πρόσδεκτε. Και επειδή Βλέπω ότι είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις ε, από τους ε, αδερφούς μου. για την ε, από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία δεν υπάρχει περίπτωση να του πάρουμε χρήματα κομπέλια. Υπάρχει αυτή η ανησυχία και μάλλον πρέπει να δώσουμε κάποιε συνεντεύξει στι εφημερίδε. Είναι πρόβλημα ότι οι λογαριασμοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Το χρήμα υπάρχει, δεν έχει χαθεί ούτε λεπτό του ευρώ. Ε, υπάρχει το χρήμα, αλλά σα παρακαλώ δαπανίστε το σωστά και με τρόπο που να επιτρέπει τη σωστή λογοδοσία. Δώστε μου να σα πληρώσω. Παρακαλώ θερμά. Διότι αν δεν πληρώνετε θα τεθεί πάλι αυτή η ερώτηση νομίζω το είπε και ο κ. ότι τι θα γίνει με τις καθυστερημένες πληρωμές. Ε, έχουμε μειώσει τις καθυστερήσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και μέχρι το τέλο τη χρονιά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν θα έχουμε καταφέρει τα πάντα όπω προβλέπαμε, αλλά παρακολουθούμε την εξέλιξη. Και αν δεν επιταχυνθεί η εκτέλεση των προγραμμάτων, ο διάδοχό μου θα χτυπήσει στο ίδιο παγόβουνο, στον ίδιο ύφαλο του backlog. Εκεί θα καταλήξουμε πάλι και θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν ε, ξεχνώ ότι αν δεν μιλήσουμε για τον Brexit δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι. Ανέκυψε σε μια-δυο παρεμβάσεις. Εδώ, ε, αυτή είναι η απάντησή μου. Βράχει πρόθεσμα. Για όσο διάστημα μπορούμε να δούμε μπροστά μα. Δεν θα υπάρξει αλλαγή. Τα δικαιώματα και υποχρεώσει ω προ τον προπολογισμό παραμένουν βάσει των εκτόσεων, βάσει των πληρωμών προ τον Βασίλειο και μετά θα πρέπει να δούμε πρώτον τι θα πει το Ηνωμένο Βασίλειο για το πού θέλουν να είναι και μετά ποιε θα είναι οι δημοσιονομικέ επιπλοκέ. Μετά θα υποδεχτούμε και μετά θα δούμε τι αποτέλεσμα θα αποφάσουμε. Ελπίζω να βρεθούμε στο σωστό σημείο. Το σωστό σημείο είναι, ελπίζω, ακόμη και σε δύσκολη θέση, να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ε, κάνω καθόλου προβλέψεις αν θα είναι λιγότερο το χρήμα, τι θα κάνουμε αν είναι λιγότερο το χρήμα, διότι απλώς δεν γνωρίζουμε τι μοντέλο θα προτιμήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και ποιε θα είναι οι δημοσιονομικέ επιπλοκέ. Όμω μπορώ να σα πω ότι δεν ε, καθόμαστε δρανεί. Εργαζόμαστε, να η ομάδα των συνεργατών μου, τα σκεφτόμαστε διαρκώ, τα μελετούμε, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει και να μα πει. Θέλουμε να κάνουμε το εξή. Και τότε θα φτάσει η στιγμή για τι διαπραγματεύσει. Σίγουρα δεν απάντησα σε όλα τα σημεία, α για το εύση ναι. Είναι διαφανές ή όχι. Εμείς ε, πραγματικά περιμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που θα μας διαφωτίσει σίγουρα για το εύση. Τα διδάγματα τα οποία έχουμε αντλήσει μέχρι στιγμής από το ΕΦΣΥ είναι ότι οι πιο προηγμένες οικονομίες και αγορές εποφελούνται όλο και πιο γρήγορα και πιο πλήρως από το ΕΦΣΥ. Αυτό προφανώς θα πρέπει να διορθωθεί με συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τις μειονεκτούσες περιφέρειες και περιοχές και θέλουμε να δούμε στις περιοχές αυτές να χρησιμοποιείται περισσότερο το ΕΦΣΥ. Στο επόμενο στάδιο θα ασχοληθούμε περισσότερο με την ενεργειακή αποδοτικότητα, με την κλιματική αλλαγή και ελπίζουμε ότι επενδύοντας τους τομείς αυτούς θα καταφέρουμε σε ένα μεταγενέστερο πιο όριμο στάδιο να έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα από το ΕΦΣΥ για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε επίσης να κάνουμε όλες αυτές τις μελέτες στις οποίες αναφερθήκατε για να δούμε αν όντως εποφελούμε θα επαρκώς από τον κοινοτικό προπολογισμό. Έχουμε ένα 20% αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιείται από τον κοινωνικό προπολογισμό για την ενσωμάτωση της διάστασης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια του κοινωνικού προπολογισμού και ελπίζουμε ότι μέσω του προγράμματος ορίζοντας 2020 θα αυξήσουμε αυτό το 20%. Περισσότερη έρευνα, περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα, μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όσον αφορά την Αφρική, Όσο πιο ελκυστική γίνεται τελικά η Αφρική για τους Ευρωπαίους επενδυτές, τόσο περισσότεροι θα είναι και οι Ευρωπαίοι επενδυτές σε αυτή την Ήπειρο. Έχουμε χάσει έδαφος ως Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μόνο μέσω της επίσημης αντιξιακής βοήθειας. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή είναι πιο ανταγωνιστικοί, κερδίζουν πολύ μεγάλα συμβόλαια στην Αφρική. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον για τους Ευρωπαίους επενδυτές στην Αφρική. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν και τις εγγύσει αυτές, τις οποίες έχουμε ήδη στα πλαίσια του προπολογισμού. Θα ήθελα να ολοκληρώσω στο σημείο αυτό, θα επανέλθω βέβαια και αργότερα, να ολοκληρώσω με δύο σημαντικά σημεία. Πρώτον, αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Σαρβαμά, ότι δηλαδή θα πρέπει να εργαστούμε έχοντας απότερο στόχο την επιτυχία. Και επιτυχία τι σημαίνει να θέσουμε τις σωστές προσδοκίες. Και τι σημαίνει αυτό, να έχουμε τον απαραίτητο συνδυασμό φιλοδοξίας αλλά και ρεαλισμού. Γιατί αν χάσουμε την υποστήριξη του Συμβουλίου, τότε αυτό το οποίο θα έχουμε θα είναι απλώς μία επανεξέταση θα έχουμε μόνο μία επανεξέταση και αυτό βέβαια δεν θα είναι θετικό. Δεν θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε το revision, την αναθεώρηση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά την απλούστευση, σα οικετεύω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε πραγματικά μία επιτροπή η οποία θα μας βοηθάει. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε αρμοδιότητες σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτό θα είναι καταγερματισμός και ουσιαστικά θα περιπλέξει τα πράγματα. Σας το ζητώ ολόψυχα λοιπόν και το ίδιο έχω πει και στο Συμβούλιο. Βέβαια όλες οι απόψεις μπορούν να ακουστούν, αλλά να περνάνε από μία μόνο επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε για την ε, παρουσίασή μου αυτή. Δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε αν παρέλειψα κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχει κάτι που δεν κάλυψα, το οποίο θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδες πρόεδρος. Ναι, η δυνατότητα που θα μπορούσε να δοθεί σε ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία δεν εξαντλούν την δυνατότητα χρησιμοποίησης των κονδυλίων συνοχής αυτά τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αποφεληθούν από κάποια άλλα προγράμματα όπως ο Ορίζοντας 2020, το Εράσμους η διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη και το καθεξή. Να σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκιο. Όντω, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να δούνε ποια είναι τα κονδύλια που έχουν στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή και στα πλαίσια τη κοινή γεωργική πολιτική και να δούμε εκεί πέρα θα μπορούσαν να τεθούν πολύ διαφορετικοί στόχοι. Τι σημαίνει αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρήματα για να πετύχουμε ένα στόχο πολιτική συνοχή ή και έναν στόχο που μπορεί να υπάγεται στον ορίζοντα 2020 ή στη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη. Πρέπει να καταρρύψουμε τους φραγμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τον έναν τομέα στον άλλον, στα πλαίσια του προπολογισμού και να υπάρχει καλύτερο συνδυασμός των κονδυλίων. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και στα πλαίσια του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ήδη από τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε το μελλοντικό πλαίσιο πολύ δύσκολα ερωτήματα έχουμε μπροστά μα αυτή τη στιγμή. Θα καταφέρουμε να δώσουμε μία απάντηση, μόνο να έχουμε ήδη από τώρα μία ειλικρινή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Φερνάντες, για 30 δευτερόλεπτα έχει το λόγο. Μία ερώτηση προς την Επίτροπο. Δεν ξέρω αν με ακούτε αυτή τη στιγμή, μιλάω γαλλικά. Καταλαβαίνω λίγο τα γαλλικά, λέει Επίτροπος. Ωραία. Η απλούστευση. Απλούστευση από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σαφώ, συμφωνώ, να έχετε έναν συνομιλητή. Τι σημαίνει όμω αυτό στην πράξη. Θα έχουμε και χαρμόσυνα νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΕΦΣΥ, ο σχετικός κανονισμός, θα έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν συνομιλητή για όλα αυτά τα ζητήματα. Κυρία Γκρέσλε, όντω συμφωνεί και αυτή ότι πρέπει να πλουστεύσουμε τα πράγματα και ιδίω να πλουστεύσουμε το δημοσιονομικό κανονισμό. Η Επίτροπος. Ναι, ναι, συμφωνώ για τα όσα είπατε για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Χρειάζεται και εκεί πέρα πλούστευση. Ο άνθρωπός μου, Νάτος, ο Ολιβιέ, εκεί πέρα είναι. Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα τα, ταλαντούχος, πολύ εργατικός, πολύ δημιουργικός. <laughs> Βάζω τελεία εκεί. Αυτός ήταν ο συνομιλητής. Ναι, ναι συμφωνούμε με τον στόχο του κανονισμού που εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ένα πουλάκι όμως μου λέει ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά και αυτές έρχονται πολλές φορές και περιπλέκουν τα πράγματα. Ότι εμπλέκονται δηλαδή στο δημοσιονομικό κανονισμό πολλές διαφορετικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήπως και εσείς πρέπει να ξεκαθαρίσετε λίγο τα πράγματα και τον τρόπο που συμβάλλετε δεν ξέρω αν οι συνεισηγητέ Όλμπρεχτ και Τωμά θέλουν να πάρουν το λόγο, ούτε ο κύριο Όλμπρεχτ ούτε η κυρία Τωμά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ κυρία Γεωργίευα. Η παρουσίασή σας πραγματικά μας επιτρέπει Εράσμους. Μας δίνεται η εντύπωση ότι είναι πάντα διαθέσιμα, αλλά όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους εθνικούς ε, αρμόδιους φορείς, μας λένε ότι σε σχέση με την αποτίμηση που γίνεται από εσά, τελικά μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στο ίμιση των κονδυλίων. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες και τους ρωτάμε τι είναι για εσά η Ευρώπη, οι περισσότεροι μας απαντούν «Για μένα Ευρώπη σημαίνει Εράσμους». Επομένως μην υποτιμάτε τη σημασία του προγράμματος αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Έχουμε κάποια σημεία ακόμα στην ημερήσια διάταξη. Είχαμε λοιπόν τις μεγάλες γραμμές του σχεδίου. Ε, προπολογισμού, ο κύριος Εστεβάν Κονσάλες Φούξ θα μας μιλήσει για την έκθεσή του. Για το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σχέδιο εκθέσεως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την Σουηδική ε, επιχείρηση Ericsson το Μάρτιο του 2016 κατέθεσε τη σχετική πρόταση η κυβέρνηση της Σουηδίας για την προστασία των 1556 εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την κινητικότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 3.250.918 ευρώ, ένα ποσοστό σημαντικό σε σχέση με τις προτάσεις Πρόκειται λοιπόν για ένα ποσό το οποίο μπορεί να στηρίξει 900 εργαζομένους με μια σειρά μέτρων που μπορούν να διευκολύνουν την επανένταξή του στην αγορά εργασίας κατόπιν εξετάσεως της προτάσεως Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στην έγκρισή της στις 5 Σεπτεμβρίου του 2016 λέγοντας ότι θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητικότητας του Ταμείου για να ενεργοποιηθεί ε, ο λόγος από όλες ήταν το συνολικό κλείσιμο της γραμμής παραγωγής σε διάφορες περιοχές της Σουηδίας και των σχετικών εγκαταστάσεων παραγωγής. Η Σουηδία λοιπόν βρέθηκε, η Έριξον συγκεκριμένα βρέθηκε συνέδεια κατάσταση λόγω της ε, οικονομικής κρίσης και του πολύ σημαντικού ανταγωνισμού πλευράς παραγωγών ε, από ασχετικά κράτη. Η επιχείρηση μείωσε σταδιακά την παραγωγή του υλικού, του hardware και οι εργαζόμενοι που έχουν χάσει τον αριθμό, το, τη θέση εργασία του παρουσιάζουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή σχετικά μεγάλη ηλικία και δεν έχουν πιθανότητε για εξεύρεση νέα απασχόληση στην αγορά. Επίσης η υποστήριξη που αποφασίζει η Σουηδική κυβέρνηση θα συμπληρώσουν τα σχετικά κονδύλια. Η Σουηδία θέλει να κατευθύνει την ε, ε, βοήθεια αυτή που θα δοθεί έτσι ώστε να ε, αναλυφθούν τα μέτρα. Το Ταμείο δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τις υποχρεώσεις της ε, επιχείρησης, όπως αυτές απορρέουν από την Εθνική Νομοθεσία, από τις λογικές συμβάσεις ή άλλα μέτρα ε, ε, σχετικά με την επιχείρηση και τον τομέα. Το αίτημα της Σουηδίας καλύπτει τις προϋποθέσεις του Ταμείου και πιστεύουμε ως εκ τούτου ότι θα πρέπει να εγκριθεί η κινητοποίηση του σχετικού ποσού ώστε να υποφεληθούν από τα μέτρα αυτά το ταχύτερο δυνατό οι εργαζόμενοι. Η κατάθεση των τροπολογιών προβλέπεται έως τις 16 Σεπτεμβρίου, βεβαίως, με πολύ μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ και ακούω τις προτάσεις σας. Merci, monsieur, monsieur. Σας ευχαριστώ, κύριε Σιγητά. Ερωτήσεις. Αν όχι ο κύριος Κονσάλης Πόντς σας είπε ποια είναι τα επόμενα στάδια και προθεσμίες. Για τους σκιώδεις των άλλων τμήματων του προπολογισμού 2017 θέλω να επισημάνω ότι η συνεδρία προβλεπόταν να ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Θα αρχίσει με το που θα τελειώσει η τωρινή μας συνεδρίαση. Ας μην ε, βιάζονται λοιπόν για τους διερμηνείς. Ε, η συνεδρία θα πάει έως τις 5.30. Ο κύριος Χριστοφόρου κύριο Σκύρτσο, συγγνώμη, για τα Ιόνια νησιά. Thank you, Mr. President. Um, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για τη χορήγηση χρηματοοικονομικής βοήθειας για περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμό τον Νοέμβριο του 2015 στην Ελλάδα. Τρία από τα Ιόνια νησιά επλήγησαν, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και μέρος της Ιθάκης. Με δύο νεκρούς δυστυχώς και αρκετούς τραυματίες. Εκτεταμένες δεν ήταν οι ζημιές στις υποδομές των τουριστικών αυτών νησιών. Άρα έχουμε αυτό το οποίο με τα κριτήριά μας περιγράφεται ως περιφερειακή καταστροφή και πρέπει να κινητοποιηθούν τα κονδύλια για να βοηθηθεί η περιοχή να αναπτυχθεί σε οικονομικούς όρους. Το συνολικό ποσό βοήθειας είναι 1,6 εκατομμύρια. Μέρος μικρό του συνολικού ποσού των 60 με 65 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπουν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές ως αναγκαίο. Η προτινόμενη κινητοποίηση δεν απαιτεί τροποποίηση στον προπολογισμό ή σχέδιο ε, αναθεώρηση του προπολογισμού του 2016 με βάση τα οποία ακούσαμε και νωρίτερα άλλωστε πρέπει να είμαστε αρκετά αυστηροί στη διαχείριση των ποσών του προπολογισμού εγώ προτείνω την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής σε ένδειξη και αλληλεγγύης προς τις πληγήσεις περιοχές της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Ευχόμαστε λοιπόν και στον εισηγητή μας να ληφθεί ταχαίως η απάντηση. Περνώ λοιπόν στη ψηφοφορία πρώτα για τις μεταφορές κονδυλίων ε, που θα μας προτείνει ο κ. Χωσέ Μανουέλ Φερνάνδες, εισηγητής του 2016. Δεν έχω, Πρόεδρε, μια ερώτηση. Είχα ήδη μάλιστα θίξει το ερώτημα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι παρούσα η Επιτροπή, αλλά θα το θίξω εγώ. Η Επιτροπή λοιπόν έχει κάνει μια, ένα έμβασμα αυτόνομο 89 99 εκατομμυρίων ευρώ ένα, για ένα νέο μηχανισμό κατεπίγουσας ε, βοήθεια στο πλαίσιο της Ένωσης. Αυτό είναι μέσα στα 10% έτσι. Όμως είναι ένας τρόπος να αντιπαρέλθει το κοινοβούλιο εγώ είχα πει ότι είχαμε δεχθεί αυτή τη νέα γραμμή με την ε, αρχική της διατύπωση, αρκεί να μην έθετε σε κίνδυνο το ε, σχέδιο για επανεγκατάσταση προσφύγων. Ενώ τώρα η γραμμή άμυφ ακόμα ε, συστέλλεται χωρίς να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο. Τα δε αυτόνομα εμβάσματα με δημοσιονομικές ή αλλά πάνω απ' όλα δημοσιονομικές συνέπειες για τι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και σημαντικά μάλιστα εμβάσματα ε, όπως αυτό των 99 εκατομμυρίων πρέπει να μας κοινοποιούνται πολύ νωρίτερα γιατί μπορούν να αποτελέσουν και έναν τρόπο να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός και μάλιστα ασορευτικά χωρίς να περνάει αυτή η ε, μεταβολή από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Και πολλές φορές μπορεί αυτό να γίνει και αντίθετα με βούληση και απόφαση του Κοινοβουλίου. Δύο εμβάσματα Φερρυπίν, τα οποία θα έπρεπε να έχουν περάσει από την Επιτροπή μας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έγερση αντιρρήσεων και ε, ενστάσεων από πλευρά του Κοινοβουλίου. Για, το έχω ξαναπεί λοιπόν. Και επιμένω πως το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τέτοιες αυτόνομες τέτοια ε, αυτόνομα εμβάσματα ακόμα και όταν είναι νόμιμα. Βεβαίω και συμφωνεί το Κοινοβούλιο. Αύριο θα είναι παρούσα η Επιτροπή στη συνεδρίαση τη Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Ω εκ τούτου θα θέσω στην, με την εκκίνηση των ε, συζητήσεων το θέμα αυτό. Για να απαντήσω. Α, δεν θα είναι εδώ αύριο. Δεν θα είναι εδώ αύριο. Άρα, στην προσοχή μας συνεδρίαση. Αρχάς Οκτωβρίου. Κύριε Ντεπρέ. Τα άλλα δύο τμήματα, κύριε Ντεπρέ. Δύο μικρά βάσματα, πρόεδρε. Χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Το ένα το ζητεί το ελεγκτικό συνέδριο και το άλλο ομπουτσμάν για το ελεγκτικό συνέδριο. Καταρχάς πρόκειται για μεταβάση 80.000 ευρώ από δύο γραμμές, από δύο κονδύλια προς το κονδύλιο παροχή ε, υπηρεσιών μετάφρασης. Το λέω αυτό γιατί και σε προηγούμενη συνεδρία είχα σημειώσει πως είχε ζητήσει την μεταφορά 126 εκατομμυρίων προς το κονδύλιο αυτό το ελεγκτικό συνέδριο και οι εξηγήσει που μας είχε δώσει το ελεγκτικό συνέδριο ήταν ότι ε, είχε βρεθεί αντιμέτωπο με σημαντική αύξηση αναγκών σε μετάφραση δεδομένη της αύξησης του αριθμού των ειδικών εκθέσεων που εκπονεί και νομίζω ότι υπάρχει εδώ εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου μάλιστα, ε, θα ήθελα να γνωρίσω ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή των ειδικών εκθέσεων, διότι είδα ε, ε έγγραφο του Ελεκτικού Συνεδρίου που πράγματι καταγράφει σημαντική αύξηση του αριθμού των ειδικών εκθέσεων. Εάν λοιπόν μας εξηγηθεί το θέμα αυτό δεν έχω αντίρρηση. Ο εκπρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου παρακαλώ. Έχετε την καλοσύνη. Αλλά μήπως κύριος Μάνκα πρώτα που ήθελε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν έχω αντίρρηση να υποστηρίξω την ε, πρόταση. ασφαλώ είναι πολύ σημαντική η μετάφραση. Αλλά θα ήθελα επί της αρχής να ζητήσω να μου απαντήσει το εξή το ελεκτικό συνέδριο. Πριν από 10 χρόνια το ελεκτικό συνέδριο είχε δημοσιεύσει έκθεση όπου έλεγε ότι όταν ένα όργανο χρειάζεται μετάφραση πρέπει να απευθύνεται σε άλλο όργανα για να, όργανο για να ζητεί την δική του ε, μετάφραση. Έτσι θα εξοικονομούσαμε 11 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχει αξιοποιήσει αυτό το μέσο, αυτή τη δυνατότητα το ελεγκτικό συνέδριο σε περιπτώσεις όπου καθυστερεί η μεταφραστική του δουλειά και δεν μπορεί η δική του υπηρεσία να καλύψει τις ανάγκες απευθύνεται στα άλλα θεσμικά όργανα για να στήσει τη βοήθειά τους απάντηση από το Ελεκτικό Συνόδριο. Ε, παρακαλώ για να δώσει απαντήσεις στα ερωτηματικά των κυρίων Ντεπρέ και Μάνκα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σε σχέση με την ερώτηση του κυρίου Ντεπρέ. Ετοιμάζει το πρόγραμμα εργασίας του το Ελεκτικό Συνέδριο στηριζόμενο στα προγραμματισμό το ετήσιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και βέβαια τις γνωμοδοτήσεις και τις ανάγκες που έχουν εκφραστεί από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, προκειμένου λοιπόν και για αυτόν τον σκοπό γίνεται συνεδρία του Πρόεδρου του Λεκτικού Συνεδρίου με, τον, με τη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών όπου συζητείται ε, ποια κοινοβουλευτική επιτροπή θέλει εις βάθος ανάλυση των λογαριασμών με ειδική έκθεση του Λεκτικού Συνεδρίου. Κατά την διαδικασία επίσης του, ε, τη απαλλαγή να τήσει αυτή η διαδικασία. Συχνά το Κοινοβούλιο ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ειδικέ και συγκεκριμένε ε, εκθέσει βάσει ελέγχων σε συγκεκριμένου τομεί. Το Ελεγκτικό Συνέδριο άπαξ και έχει ετοιμάσει το πρόγραμμα εργασία του, το παρουσιάζει ε, στο ελεκτικό συνέδριο και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού πάντα Ιανουάριο μήνα ώστε να βεβαιωθεί ότι και τα αιτήματα που έχουν εκφραστεί έχουν ληφθεί επαρκώ υπόψη στο πρόγραμμα εργασία του Ελληνικού Συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά την άλλη ερώτηση ως προς την ε, αμοιβεοποίηση αυτών των αναγκών σε μετάφραση. Έχουμε ζητήσει και από τις υπηρεσίες του Συμβουλίου και από αυτές τις επιτροπές να μας στηρίξουν σε μεταφραστικές ανάγκες και όντως μας έχουν ε, προσφέρει τη βοήθειά τους. Το συγκεκριμένο πόσο που ζητούμε έχει να κάνει με εξωτερικές αναθέσεις μετάφρασης για τις χώρες που έχουν γλώσσες περιορισμένης διάδοσης και για τις οποίες αναγκαζόμεθα να προσφεύγουμε σε εξωτερική ανάθεση. Ξέρετε ότι γλώσσες εκτός των γαλλικών, αγγλικών, γερμανικών έχουν πολλές φορές ε, συγκεκριμένη ανάγκη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και κατά τρόπο επίγοντα βέβαια. Ο εισηγητής παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου για την απάντησή του. Μας ξανάριξε, μας ξανάστελε το μπαλάκι αφού μέσω ημών φαίνεται έχει την έγκριση, μέσω ημών ω μέλου τη διάσκεψη των Πρόεδρων φυσικά, Ευχαριστώ. Αντίρρηση από τα μέλη της Επιτροπής υπάρχει, αφού ο κύριο Δεπρέ δεν έχει αντίρρηση. Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν το σχετικό έμβασμα. Ομπουτσμαν, Ναι, Πρόεδρε, εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Πρόκειται για έμβασμα της τάξης των 138, 138 1.900 ευρώ ε, και μας επιτρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε ανάγκες όπως την ανάπτυξη της του ιστοτόπου, κάλυψη αναγκών στο νέο αυτό το οποίο διατίθεται για τον διαμεσολαβητή και άλλα ε, μικροποσά. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αιτιολογημένο το αίτημα και ε, δεν μένει παρά να το εγκρίνουμε. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Αντιρρήσεις υπάρχουν, πάντα χωρίς μικρόφωνο. Ο πρόεδρος δεν ακούγεται. Wir Ναι, ένα θέμα έχουμε για τα κτίρια. Πάει όμως γρήγορα, θα σας τα πω όμως σύντομα. Πρόκειται για ένα κτίριο της εξωτερικής υπηρεσίας ε, στο, στη Νότιο Κορέα για τον πύργο S, S Tower πρόκειται με κάποια προβλήματα τα οποία διωγγώθηκαν σύντο χρόνο ε, δεν είχαμε αρκετό χώρο και έτσι χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι και το 12ο όροφο με τέσσερις όροφους συνολικά που καταλαμβάναμε. Μετά άρχισε η ανακαίνιση με εργασίες ε, ε, που σε ένα βαθμό οφείλονται και στο γεγονό ότι και άλλα κράτη-μέλη άρχισαν να ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτές τις εργασίες. Κόστος σε σχέση με το παλαιό κτίριο είναι ελαφρώς χαμηλότερο το κόστος του νέου κτιρίου, ουσιαστικά όμως το ίδιο, με περισσότερο χώρο όμως, με περισσότερους κοινού χώρους επίσης. Λετωνία και εσθονία θα καλύπτονται από τους χώρους αυτούς μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι είναι και η Φιλανδία και η Δανία επίσης έτοιμες να εγκατασταθούν. Καλά λέει ο κύριος Δεπρέ, ναι, πολύ ωραία. Στο ίδιο κτίριο. Ναι και δεν με θέλει να ακούσει ο Ζεράρ και μάλλον ε, προτιμά να φύγει από εδώ. Ε, πιστεύω ότι αν δεν έχουν συναδέλφοι άλλες αντιρρήσεις, τα έχω επαληθεύσει ε, όλα το συνολικό κόστος λοιπόν ανά ε, τόσο. Έχουμε συνολικά 1,6 ε, εκατομμύρια και 765.000 για την αναμόρφωση, Επομένω δεν είναι πολύ ψηλά τα ποσά και νομίζω ότι μπορούμε να το εγκρίνουμε. Αν δεν έχει αντίρρηση ο πρόεδρος, ας το εγκρίνουμε λοιπόν. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχω Είχα ακούσει κάτι φήμες ότι θέλατε να καθυστερήσετε λίγο για να λάβετε πιο πολλές πληροφορίες. Εσείς μας λέτε τώρα ότι έχετε κάνει την ανάλυση και άρα μπορούμε να το εγκρίνουμε. Ναι, η ΕΑΕ είχε αρχικά δώσει περιορισμένες πληροφορίες που μας φάνηκαν κάπως υπερβολικές. Τους υποδείξαμε ότι είχαν μάλλον κάνει λάθος τους υπολογισμούς τους κατά 3 εκατομμύρια και βεβαίως το διόρθωσαν με πολύ φιλική συνεργασία και ύφος. Αν και μου κάνει εντύπωση ότι έκανε λάθος της τάξεις των 3 εκατομμυρίων στους λογαριασμούς της. Ελπίζω στο μέλλον να μην ε, επαναληφθεί. Αλλά πάντως δεν υπάρχει πρόβλημα σχέση με τα, με τα τωρινά στοιχεία. Καλώς λέει ο πρόεδρος Τρία εκατομμύρια λαφάκι είπατε. εν πάση περιπτώσει σε σχέση με αυτό που κόστιζε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι, προ, οι προηγούμενες εγκαταστάσεις στην Νότια Κορέα, νομίζω ότι δεν επιβαρυνόμαστε με αυτή την επιλογή με νέες ε, με νέε δαπάνε. Επομένω, πρέπει να το εγκρίσουμε. Ε, Α σηκώσουμε το χέρι. Λοιπόν, ποιο είναι υπέρ των προτάσεων του συγκητή. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχέ. Ομόφωνα, λοιπόν, εγκρίνεται. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. 9 η ώρα. Επιτροπή πάλι. Και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Πέρα συνεδριάσεως.